Ladies Κυρίες και κύριοι, ορίσατε θερμά στην ε, συγκινή συνεδρία Επιτροπής Εξωτερικών, ε, Επιτροπής Ανάπτυξης και Επιτροπής Προϋπολογισμών. Σήμερα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με εμπειρογνώμονες και ενεχομένου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης, το λεγόμενο ΕΤΒΑ παρακαλώ στα ελληνικά. Και είμαστε πάρα πολύ ε, περήφανη γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη παίζει σημαντικό ρόλο. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που βαρύνουν πολύ ε, την πολιτική μας λήψη αποφάσεων και χαιρόμαστε γι' αυτό το εγχείρημα και την άσκηση που θα κάνουμε σήμερα. Θα έχουμε μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη που μπορεί να είναι μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως. Αυτό το σχέδιο για τις εξωτερικές επενδύσεις θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο και πρωταγωνιστικό ε, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει διάφορες προσπάθειες ε, σε άλλα μέρη του κόσμου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ύπεθρος κυριαρχούν σε αυτές τις δραστηριότητες και με μεγάλη χαρά θα κάνουμε τη σημερινή συζήτηση για να δούμε πώς μπορούμε να επικεντρωθούμε για να έχουμε πιο συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα για τους πολίτες μας στην ανάπτυξη. Όπως γνωρίζετε, οι επιτροπές μας έχουν εργαστεί από την περασμένη εβδομάδα από τις 28 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα, μετά την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, παρουσία ε, του Κατάινεν και της ε, Μοντιγκερίνη οι οποίοι είναι αρμόδιοι. Ελπίζουμε να βρούμε και μια άλλη ευκαιρία να ε, κάνουμε συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα. Νομίζω αυτό είναι ο σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε. Στο μεταξύ όμως έχουμε και τους τρεις εισηγητές. Βλέπω εδώ τον κύριο Κούκαν. Καλώς ορίσατε θερμά και σας ευχαριστώ πολύ που δραστηριοποιήσετε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Επίσης, άλλος εισηγητής είναι ο κύριος Φροντσούλικα. Και χαίρομαι που βλέπω να ενδιαφέρονται οι βουλευτές για αυτά τα θέματα. Θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ενημέρωση από του συναδέλφου. Βεβαίω έχουμε και από την Επιτροπή Προπολογισμών τη συνάδελφο Αίντερ Γκάρδια Σάμπα Ρουμπιάλ. Είμαστε συνάδελφοι στην Επιτροπή Προπολογισμών. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε αγαστά και στα θέματα περιβάλλοντος, μάλλον στα θέματα ανάπτυξη στην Επιτροπή Προπολογισμών. Και μπορούμε και καλά συνεργαζόμαστε και εγκαίρω να υποβάλουμε τι εκθέσει. Το σχέδιο έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και θα συζητήσουμε στην επόμενη κοινή μας συνεδρίαση στις 21 του μηνός. Έχουμε υποβάλει και γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε λάβει τη Δευτέρα γραπτές απαντήσεις. Όλα αυτά έχουν γίνει μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Καλές ικανοποιητικές οι απαντήσεις. Και σήμερα καλέσαμε λοιπόν εμπειρογνώμονες και ειδικού για να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους, τις εμπειρίες τους για το ταμείο αυτό, τα προβλήματα και τις επιτυχίες που αναμένουμε. Και θέλουμε να ακούσουμε από εσά τι έχετε να μας πείτε, τι περιμένετε από εμά. Ξέρετε, στην πολιτική ζωή υπάρχουν διάφορες επιλογές και ο καθένας καλείται να δει πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε αποκρισταλωμένη άποψη, ούτε αιμονές, ούτε λέμε έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και δεν θέλουμε να ακούσουμε κανέναν εξωτερικό, ίσα ίσα. Γι' αυτό σας καλέσαμε και γι' αυτό θέλουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις με τους ενδιαφερομένους. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά λοιπόν, δώσουμε ε, το λόγο στου συμπροέδρους. Και χαίρομαι που είναι εδώ ο Χαβιέ Κόουσο, ε, αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΑΦΕΤ και ο Νόρμπετ Νόιζερ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Ε, Χαβιέ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, θα μιλήσω ισπανικά. Εξ ονομά της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στη σημερινή κοινή μα συνεδρίαση. Σε αυτή την ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε του ενδιαφερομένου για την πολύ σημαντική νομοθετική πρόταση. Επειδή είναι εξαιρετικά περιορισμένο ο χρόνο μα και έχουμε μακρύ κατάλογο εξεχόντων ομιλητών, θέλω να σα πω μόνο μου επιτρέπετε ότι περιμένουμε να ακούσουμε από εσά τι να κάνουμε έτσι ώστε το Ταμείο βιώσιμη ανάπτυξη, να στεφτεί με επιτυχία. Αυτό είναι ο κοινό μα στόχο θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάπτυξη και ενίσχυση των, ε, των σχέσεων με τους εταίρους, στη γειτονία και να δούμε θέματα μετανάστευσης που αντιμετωπίζουμε όλοι. Και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν οι τοποθετήσεις σας και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Νόιζερ από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ σύντομα, διότι το σημαντικότερο σήμερα είναι βεβαίως να ακούσουμε τους διαφόρους εμπειρογνώμονες, να αναπτύξουν τις ιδέες, την εμπειρία τους, τη γνώση τους για την ενασχόλησή μας με το σημαντικό αυτό νομοθέτημα. Από την εποχή που άρχισε η δημοσιονομική κρίση, οι άμεσες εξωτερικές επενδύσεις και άλλες ροές ιδιωτικών κεφαλαίων σε αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μειωθεί. Το 2012 μόνο 6%, δηλαδή 34,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το σύνολο των αλλοδαπών άμεσων επενδύσεων που γίνονται σε αναπτυσσόμενες χώρες, μόνο λοιπόν αυτό το 6% πήγε στις λεγόμενες εύθραυστες χώρες. Δηλαδή, κατά μέσον όρο επένδυση 23 ευρώ κατά κεφαλή, σε σύγκριση με τα 128 ευρώ, δηλαδή το πενταπλάσιο που επενδύονται σε άλλε αναπτυσσόμενε χώρε. Η επιτυχία λοιπόν του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμη ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από το εάν θα μπορέσει να, προωθήσει, να προωθήσει συγγνώμη, επενδύσεις σε τέτοιες χώρες που έχουν υψηλό κίνδυνο και μικρές, μικρά χαμηλά επίπεδα άμεσων επενδύσεων. Εάν αυτό επιτύχει λοιπόν θα είναι πραγματικά μια προστιθέμενη αξία. Το πόσο σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το εξήγησε πρόσφατα σε επιστολή του ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, επιστολή προς τον κύριο Ταγιάννη. Το χρονοδιάγραμμά μας είναι επίσης φιλόδοξο. Δεν επιτρέπεται ωστόσο να επιβαρύνει την ε, μελέτη του νομοθετήματος στην ουσία. Οι άνθρωποι και στην Ευρώπη αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν αρκούνται σε σύμβολα. Ούτε τους αρέσουν αυτοί οι λεγόμενοι λευκοί ελέφαντες που τέτοια παραδείγματα υπήρξαν μέχρι τώρα στην αναπτυξιακή συνεργασία. Θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα μπορέσει να αποδώσει εκεί όπου χρειάζεται. Ω Επιτροπή Αναπτύξεω γνωρίζουμε απολύτω ότι θα χρειαστούν ποσά σε ύψο δισεκατομμυρίων για να επιτευχθεί πραγματική πρόοδο σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την επίτευξη των ε, στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτά τα δισεκατομμύρια δεν θα προέλθουν μονάχα από την δημόσια χρηματοδότηση. Χρειάζεται λοιπόν μια προσέγγιση που θα προωθήσει και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε ωστόσο το αποτέλεσμα μόχλευσης και να φροντίσουμε να επενδύσουμε σε έργα τα οποία θα οδηγήσουν και σε οικονομική ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα και σε μείωση της φτώχειας και τα οποία δεν θα βλάψουν τους πτωχότερους των πτωχών, για παράδειγμα μέσω του λεγόμενου land grabbing, της αρπαγής γεών ή με αναγκαστικές μετεγκαταστάσεις, πράγματα τα οποία έχουμε δει να γίνονται από μεγάλες επενδύσεις. Για το λόγο αυτό, το Ταμείο και οι επενδύσεις είναι και ένα σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Αναπτυξιακή Πολιτική, όπου εγώ είμαι συνεισηγητής. Εκεί σώμεθα υπέρ μιας πλήρους πρόσβαση σε πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και το δικαίωμα να έχει καθεστώς παρατηρητού, διότι θέλουμε να γνωρίζουμε ότι οι εγγυήσει που προέρχονται από τις επενδύσεις θα οδηγήσουν πράγματι σε ανάπτυξη και σε βιώσιμη μείωση της φτώχειας. Θα πρέπει να προσανατολίσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολυνθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό το λέω διότι είμαι πεπισμένο ότι ιδίως οι γυναίκες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη. Πρέπει οι επενδύσεις να έχουν ένα χαρακτήρα ηθικό, κοινωνικά υπεύθυνο και βιώσιμο. Αυτό ισχύει και για τις ιδιωτικές αλλά και για τις συνεταιρικές και δημόσιες επενδύσεις που θα γίνουν δηλαδή σε αυτούς τους τομείς. Με μεγάλη περιέργεια παρα, ε, περιμένω μάλλον τις ε, προτάσεις των εισηγητών μας του σημερινού απογεύματος. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε τώρα στο πρώτο πάνελ. Πάνελ number one. Χαίρομαι πολύ που έχουμε κοντά μας τον Πρόεδρο και εκτελεστικό διαχειριστή του Ευρωαφρικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κύριο Γουαταρά, που είναι εμπειρογνώμων σε θέματα προώθησης επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε να αναμειχθούν οι επιχειρήσεις, οικογενειακές και άλλες που αποτελεί πρώτη στο στόχο μας, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να πετύχουμε να παραμείνει ο κόσμος στις περιοχές της υπαίθρου, να έχουν δηλαδή εκεί επιτυχημένες επιχειρήσεις οι οποίες θα του εξασφαλίσουν την απασχόληση. Σας αναμένουμε λοιπόν να μας εξηγήσετε τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευκαιρία που μας δίνετε. Να σα θυμίσω, πρόκειται για ένα εμπορικό επιμελητήριο που είναι εγκατεστημένο στι Βρυξέλλες εδώ και λίγο παραπάνω από τέσσερα χρόνια. Εργαζόμαστε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα στην Αφρική και στην Ευρώπη μέσα σε μια προοπτική βιώσιμη ανάπτυξη. Για κάποια χρόνια διοργανώσαμε εκδηλώσει όπου ήρθαν σε επαφή αυτοί οι φορεί και έχουν ανταλλάξει απόψει και εδώ και δύο χρόνια συνειδητοποιήσαμε ότι χρειάζονταν κάτι παραπάνω από τι ανταλλαγέ απόψεων και τι συζητήσει. και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα πρόγραμμα που λέγεται Access Fin και έχει στόχο την διευκόλυνση της ε, πρόσβασης στη χρηματοδότηση στον επιχειρηματικό τομέα. Ε, έχουμε επίσης σημαντήσει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο ε, και ακριβώς η ευκαιρία η σημερινή είναι απόλυτα επίκαιρη. Να σας πω λοιπόν πώς βλέπουμε εμείς ε, τα πράγματα επιτόπου όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τον ιδιωτικό τομέα στην Αφρική. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε τρεις κατηγορίες. Έχουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε τους επιχειρηματίες και ε, τον ε, τομέα της... τον άτυπο. Ε, αυτοί είναι οι τρει βασικοί τομείς. Ε, οι επιχειρήσεις που όμως χρειάζονται χρηματοδότηση συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν ε, ευκαιρίες εμπορικές και τις οποίες όμως χρειάζονται χρηματοδότηση, χρειάζονται κονδύλια. Όμως αυτές οι εμπορικές ευκαιρίες είναι περιορισμένες χρονικές διάρκειες, δύο-τρεις μήνες. Δηλαδή πρόκειται για συμβάσεις που πρέπει να αρχίσουν να εκτελούν. Και άρα η διαδικασία συλλογή κονδυλίων είναι πιο μακρά από την διάρκεια εκτέλεση των συμβάσεων, τουλάχιστον Δυτική Αφρική, την οποία γνωρίζω αρκετά καλά, το πρόβλημα είναι η οι προθεσμίες πρόσβασης στην χρηματοδότηση εγγύησης που ζητώνται από τις τράπεζες και συνειδητοποιούμε τελικά ότι υπάρχει πρόβλημα όχι όσον αφορά τις ε, δεξιότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ε, το θέμα είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν επί τόπου και να παρακολουθήσουν ε, τις επενδύσεις. Δίνουν τα κονδύλια μόνο εκεί που υπάρχει απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν χρειάζονται τέτοιου είδους συμμετοδότηση Χρειάζεται ενίσχυση δυνατοτήτων στο management, στο ανάπτυξη την επιχειρηματική. Γι' αυτό χρειάζεται συνοδεία και ε, συμπαράσταση επιτόπου. Γι' ε, αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Να έχουμε δηλαδή ανθρώπου ε, οι οποίοι θα ανασκουμποθούν, θα πάνε επιτόπου και θα συνεργαστούν στενά με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο λοιπόν που πρέπει να εντοπιστεί. Και το δεύτερο που μπορούμε να αναφέρουμε είναι οι εγγυήσει. Οι εγγυήσει είναι υπερβολικέ. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα που συνέβη πολύ πρόσφατα. Μια επιχείρηση που χρειαζόταν να να αγοράσει ε, ε, εξοπλισμό μεταφορών, δηλαδή ε, μεγάλα μηχανήματα και φορτηγά για συνεργασία με ένα ορυχείο. Ζήτησε λοιπόν εγγύηση η τράπεζα, έδωσε ως εγγύηση η επιχείρηση τα μηχανήματα και τα φορτηγά που ήθελε να αγοράσει και άρα η τράπεζα είχε καταρχάς την εγγύηση που χρειαζόταν. Εμείς συνομιλήσαμε με την τράπεζα, τα είχαμε όλα διοργανώσει και την τελευταία στιγμή η τράπεζα ζητά λοιπόν, απαιτεί μάλλον, να υπάρχουν και διαθέσιμα χρήματα στο λογαριασμό της επιχείρησης πριν να καταβάλει τη κοντήλια. Ενώ έχει ήδη ε, τις, ε, το λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας, δηλαδή είναι ε, υπερβολικές εγγύησεις που απαιτεί η τράπεζα. Εκεί είναι απλά ένα παράδειγμα. Άλλος ε, κοινό στόχος είναι ήδη οι επιχειρηματίες γιατί οι περισσότεροι μηχανισμοί εγγυήσεων αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνονται στα projects των επιχειρηματιών. Απαιτείται και απαιτώνται καινοτόμα σχέδια. Πρόκειται για ένα ή δύο εκατομμύρια δολάρια ως μίνιμουμ οι επιχειρηματίε δεν έχουν τέτοιου είδους κονδύλια. Είναι καλό να μιλάμε για καινοτομία, αλλά υπάρχουν πράγματα βασικά, βασικές υπηρεσίες που δεν υπάρχουν και που μπορεί να απασχολήσουν και κόσμο τοπικά. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει αυτός ο στόχος όσον αφορά τι επιχειρήσεις. Τελευταία μου παρατήρηση αφορά τον άτυπο τομέα, ο οποίος ε, ε, χειρίζεται πολλά χρήματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μετρώνται πουθενά αυτά γιατί φοβούνται το η φορολογία, δεν θέλουν αναορατές δραστηριότητε. Υπάρχει δηλαδή ε, ε, μεγάλη παραοικονομία. Το εμπόδιο όμως είναι ότι πολλοί δεν είναι καν μορφωμένοι, δεν ξέρουν πώς να χειριστούν την οικονομία. Έχουν χρήματα μετρητά που δεν ξέρουν να τα τοποθετήσουν, ούτε να τα βάλουν στην τράπεζα. Πρέπει και εκεί λοιπόν να υπάρξει ε, συμβουλευτική δραστηριότητα για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια της παραοικονομίας. τώρα, από την εμπειρία μας και προς αυτή την κατεύθυνση κατευθυνόμαστε και ε, γι' αυτό και καλούμε τους εταίρους μας να έρθουν κοντά μας. Ε, ε, είναι βασικό να πάμε επί τόπου να εντοπίσουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά μην αρκεστούμε στο να του χρηματοδοτήσουμε, αλλά να του συνοδεύσουμε σε αυτήν τη χρηματοδότηση. Και αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουν δοθεί τα χρήματα, να μπορούμε να τους βοηθήσουμε στη διαχείριση στις δαπάνες, στα έσοδα για μια κάποια περίοδο, ώστε πραγματικά να εξασφαλίσουμε μέσω coaching και ενίσχυση των δυνατοτήτων ότι έχουν τη δυνατότητα και τις σωστές ε, ε, συμπεριφορές. Κάτι ακόμα θα ήταν με τις τοπικές τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τοπικά να υπάρχει ε, συνεργασία. Να σας δώσω το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που δίνει χρήματα σε κάποιες τράπεζες. Δεν λειτουργεί πολύ καλά το σύστημα γιατί αυτές οι τράπεζες τα προσθέτουν στο σύνολο των πόρων που έχουν και τις διαχειρίζονται όπως ε, συνηθίζουν. Δηλαδή αποφασίζουμε σε ποιον θα έπρεπε να δοθεί κάποια πίστοση ή όχι επί τη βάση ανάλυσης κινδύνου και κάλυψης ε, εγγύσεων. Μια λύση που μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα είναι να μείνουν αυτές οι τράπεζες ως φορείς που θα λαμβάνουν τα χρήματα, αλλά να υπάρχει και ένα τρίτο φορέας ο οποίο ακριβώς εκείνος θα είναι που θα λάβει την απόφαση να αναλύσει την αίτηση πίστοση και να χορηγήσει τη χρηματοδότηση ή όχι. Δηλαδή η τράπεζα έτσι να μπορεί να παίξει το ρόλο της γιατί η νομοθεσία ζητά κάποιες ζητα καποιες εγγυήσει για να υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπορεί να δώσει χρήματα, αλλά ε, να είναι υπεύθυνη ε, επί τη βάση ε, όμως ε, της κρίσης αυτού του τρίτου μέρος του τρίτου οργανισμού. Πιστεύουμε πως ε, κάτι τέτοιο θα μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει. Σε αυτά λοιπόν θα σταματήσω και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Yes, many things. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρόμαστε να ακούμε κάποιον που έχει εμπειρία επιτόπου ε, δηλαδή ε, που ξέρει αυτά που αποφασίζουμε πώς γίνονται δεκτά στο άλλο άκρο και τι θέλει ο κόσμος εκεί και τι περιμένει από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια αυτά. Ακολουθεί η κυρία Αλίσα Χίθ ε, από το PRI, αρχές για υπεύθυνη επένδυση. Senior Policy Manager. Καλώς ορίσατε και σας παρακαλούμε να μοιραστείτε και εσείς μαζί μας τις ιδέες και τις εμπειρίες σας. Ευχαριστώ. Μου ζήτησαν να πω δύο πράγματα σήμερα. Πρώτον, να σας συστήσω την οργάνωσή μας, το PRI, και ε, δεύτερον, να δούμε πώς συνδέονται οι επενδύσεις με την ανισότητα. Αρχίζω πολύ γρήγορα οργάνωσή μου που λέγεται Principles for Responsible Investment έχουμε συσταθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ε, είμαστε ένας ανεξάρτητος ε, φορέας που βοηθάει στη λήψη των αποφάσεων της κυβερνήσεις και τους ενδιαφερομένους. Αυτό έχει να κάνει και με την ε, ευρύτερη οικονομία, τη σταθερότητα της 1.700 ε, έχουμε ε, ως μέλη, οι περισσότεροι στην Ευρώπη με ένα τεράστιο κύκλο εργασιών. Οι περισσότεροι είναι ε, ειδικοί στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων και των κρατών. Οι περισσότεροι όμως είναι από εταιρείε ασφαλιστικές και παιδιτικές. Δεν είναι η δικότητά μας οι επενδύσεις στην ανάπτυξη, αλλά κάποια από τα σημεία που συζητούμε σήμερα ε, μας αφορούν και έχουν να κάνουν με τη δική μας δραστηριότητα. Αρχίζω λοιπόν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ε, για τους ε, στόχους του Ταμείου. Δεν μπορεί να έχει κανείς ένα εξαντλητικό κίνδυνο των ε, κινδύνων και των ευκαιριών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ταμείο. Μια στιγμή γιατί έχω και κάτι διαφάνειες ξέχασα. Η χρηματοδότηση μιας επένδυσης εξαρτάται από πολλά πράγματα, από την νομοθεσία, από το πώς γίνεται μια δημόσια συζήτηση ε, για προβληματικές συμπεριφορές, για προβληματικές επενδύσεις και ποια είναι η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Αντί να φτιάξουμε ένα κατάλογο, ε, εμείς λέμε οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν μια διαδικασία για να καταλάβουν την πραγματικότητα της κάθε χώρας και τι συμβαίνει όταν γίνεται μια επένδυση. Κάθε χρόνο ε, συμβουλευόμαστε τα μέλη μας και μαθαίνουμε από τις εμπειρίες τους. Υπάρχουν κάποια διεθνή στάνταρ και προδιαγραφές ε, που έχουν να κάνουν με την επένδυση διεθνώς. Τι ισχύει, ποιες είναι οι πρακτικές, οι επιχειρηματικές, τι θεωρείται παραδεκτό και τι απαράδεκτο. Υπάρχουν οι παγκόσμιες αρχές του ΟΗΕ σε πολύ ψηλό επίπεδο Υπάρχει ε, οι συμβάσει του ε, ILO, η Οικουμενική Διακήρυξη των ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Σύμβαση κατά της Διαφθοράς των Ηνωμένων Εθνών και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ για τις πολυεθνικές. Όλα αυτά εστιάζουν στην οικονομία. Όταν μιλούμε όμως για επενδύσεις σε αναδυόμενες οικονομίες, είναι πολύ λιγότερο διαρθρωμένα τα πράγματα και οι επενδυτικές εταιρείε δεν αποκαλύπτουν και πάρα πολλά στοιχεία. Δεν ισχύουν ε, όλα αυτά τα πολύ θεωρητικά παντού. Υπάρχουν και κάποια περιβαλλοντικά πρότυπα και προδιαγραφές και κοινωνικά επίσης. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που είναι τεράστιο κεφάλαιο ε, στην επενδυτική κοινότητα που κάνει υπεύθυνε επενδύσεις και πώς ανταποκρίνονται τα μέλη μας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ε, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, τι επιπτώσεις έχουν στις επενδύσεις. Μερικοί είναι πολύ πιο εύκολοι να χρηματοδοτηθούν και άλλοι λιγότερο. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ποια επένδυση εντάσσεται στους βιώσιμους στόχους. Υπάρχουν κάποιες αρχές για ε, θετική χρηματοδότηση με θετικό αντίκτυπο που μπορούν οι επενδυτές να αναλύουν και να εξηγούν ε, ποια είναι η περιβαλλοντική, κοινωνική και γενικότερη επίπτωση των επενδύσεων τους. Έρχομαι τώρα στην ανισότητα. Θα πρέπει οι επενδυτές να το προσέξουν αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, η ανισότητα στο εισόδημα μπορεί να σημαίνει αστάθεια ε, και πρόβλημα σε μια οικονομία, οπότε δεν θα έχει μακροπρόθεσμη μια απόδοση, μια επένδυση. Και επίσης ε, ε, επηρεάζει και το γενικότερο περιβάλλον, είναι ανησυχία και κυριαρχεί στη συζήτηση σε πολλές χώρες, άρα αυτό μπορεί να είναι ένα εμπόδιο για την επένδυση. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω τις προσεγγίσεις των μελών μας σε σχέση με αυτό. η ανισότητα χρησιμοποιείται ως ένα πρίσμα για, την ανάλυση μιας επένδυσης. Αυτό είναι μια σχετικά νέα ιδέα. Τι έχουμε διαπιστώσει όμως, με πρακτική ετών για ε, ε, υπεύθυνε επενδύσεις υπάρχουν κάποια θέματα ε, στα οποία εστιάσαμε που συνδέονται με την ανισότητα στο εισόδημα. Σας δώσω κάποια παράδειγμα. Πόσο απέχει η αμοιβή ενός στελέχους μιας εταιρείας από έναν αδικευτό εργάτη, ε, να υπάρχουν ε, δείκτες όπως η σταθερή απασχόληση, η απόδοση και η εργασία να αναγνωρίζεται ως δημιουργία υπεραξίας και όχι απλώς ε, ένα έξοδο για τον επενδυτή, το μισθολογικό κόστος εργασίας δηλαδή. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες ε, όπως είναι η χαμηλή μισθή, η έλλειψη ε, σταθερών προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής συνεργασία. Πολλές φορές οι επενδυτές δεν θέλουν να συνδέουν το όνομά τους με τέτοιες καταστάσεις. Και επίσης υπάρχουν και ανισότητες ε, εισοδήματος στις χώρες που είναι κίνδυνος αποσταθεροποίησης και πολιτικής αποσταθεροποίησης ενός κράτους και κάθε φορά που αναλύει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες μιας επένδυσης πρέπει να λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να σας αναφέρω είναι ε, στοχευμένες επενδύσεις για να μειωθούν οι ανισότητες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοια παραδείγματα σε κάποιες χώρες ε, με παραδοσιακούς ε, στόχους σε επενδύσεις ε, στη στέγαση ή στην παροχή, παραγωγή μάλλον ενέργειας. Ε, άλλο θέμα που θέλω να σας αναφέρω είναι ε, η αντιστροφή της πυραμίδας, δηλαδή θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες και αγαθά στα πιο φτωχά στρώματα της κοινωνίας. Έχουμε βρει ότι πολλοί θεσμικοί επενδυτές, ιδιαίτερα εκείνοι που συνδέονται με την εργασία, έχουν αρχίσει να βάζουν πολιτικές για υπεύθυνες συμβάσεις, στην υπογραφή της σύμβαση, ιδιαίτερα ε, με ταμεία διαρθρωτικά, με ταμεία για την πρόσβαση στην κτηματαγορά για, και θέτουν ως προϋπόθεση τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις για να γίνει καν επένδυση. Ε, αν θέλετε μπορούμε στη συνέχεια να επεκταθούμε και να απαντήσω και σε ερωτήσεις. Yes, first of all, thank you so much. σας ευχαριστούμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ που παραμείνατε και μέσα στο χρονικό όριο που σας είχαμε διαθέσει. Αυτό είναι καλό διότι έτσι θα έχουν την ευκαιρία όλοι να μπορέσουν να ομιλήσουν και να προχωρήσουμε τώρα στον επόμενο ομιλητή που είναι ανώτατος αξιωματούχος του Development Policy Management ο κύριος Σαν Μπιλάλ. μεγάλη χαρά τον έχω κοντά μου. Γνωρίζουμε ότι ο οργανισμός του παίζει πολύ κέριο ρόλο και πολύ ευχαρίστως ακούμε τις συμβουλές του. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Εμεί είμαστε ένα είδο think and do tank, δηλαδή δεξαμενή σκέψη και πράξη. Για την συνάντησή σα, μου ζητήθηκε να σα πω ορισμένα πράγματα για το blending, για την ανάμειξη δηλαδή των διαφόρων μορφών χρηματοδότηση. Μια στιγμή να δω αν λειτουργεί ε, ο τηλεχειρισμός για τις διαφάνειες. Έχω κάποιε διαφάνειες, αλλά τέλος πάντων. Ε, θα ήθελα τώρα να, προ, να πω πρώτα ότι αυτή, αυτό το blending, αυτή η σύμμιξη είναι μια από τις μορφές που χρησιμοποιεί το EFSD, το Ευρωπαϊκό Ταμείο δηλαδή Ανάπτυξη, Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης, γιατί ορισμένες φορές ακούμε σε ομιλίες, ιδίως σε κύκλους των Βρυξελών και μεταξύ αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι το blending ε, δεν ικανοποιεί. Αλλά δεν είναι και καμιά πανάκια, είναι ένα από τα πολλά συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποφευθούν, για παράδειγμα, και ε, μη νόμιμες επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις, στρέβλωση της αγοράς κλπ. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το blending να θεωρηθεί ως ένα από τα εργαλεία που έχει η διεθνής κοινότητα στην ε, διαθεσή της για να δώσει λύσεις. Όταν εξετάζουμε την σύμμιξη αυτή, το blending, υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί. Και γίνονται συζητήσεις στο διεθνές επίπεδο μεταξύ των διαφόρων ε, τραπεζών αναπτύξεως να σκεφτούμε, να βρούμε ένα κοινό ορισμό. Γιατί αυτό το blending που χρησιμοποιούμε βασίζεται σε διαφορετικούς ορισμούς. Κάτι το οποίο οδηγεί σε ένα κατακαιρματισμό. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη συνέπεια και συνέχεια στον ορισμό και στους ορισμούς και πιο πολλές κοινέ αρχές και τρόποι εφαρμογής για το blending. Τώρα τα υπέρ και τα κατά. Υπάρχουν πολλά υπέρ του blending, αφενός δηλαδή ότι δίνει ε, μια μόχλευση, δηλαδή μπορεί να επιτύχει κανείς περισσότερα πράγματα με λιγότερα χρήματα, με λιγότερους πόρους επιτρέπει την μόχλευση πολλών περισσότερων πόρων. Έχουμε και την Ατζέντα 2030 και τη χρηματοδότησή της που βοηθεί να κλείσουν τα χρηματοδοτικά κενά. Έχει λοιπόν μια ελκυστικότητα και σε ό,τι αφορά την ποιοτική χρηματοδότηση αλλά και την ποσότητα. Εξετάζοντας κανείς τα θετικά, θα κάνει μια σύγκριση, έτσι. Δηλαδή είναι καλύτερο σε σχέση με τι. Είναι προτιμότερο από την ε, παραδοσιακή επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι καλύτερο από την βοήθεια που δίνουν ε, τα Ιδρύματα Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης. Χρειάζεται δηλαδή σύγκριση με ε, κάποια άλλα, με κάποιους άλλους θεσμούς. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και σε ό,τι αφορά και τις αρνητικές πτυχές του. Ε, το blending, αυτή η ανάμειξη, δεν είναι βέβαια για όλες τις προκλήσεις. Υπάρχει ο κίνδυνος να ανατραπούν κάποιες ε, αρχές της χρηματοδότησης, να αντικατασταθούν οι ιδιωτικοί πόροι από τα χρήματα αυτά αντί να μοχλευτούν. Υπάρχει ενδεχόμενα πρόβλημα και με την προσθετικότητα, εφόσον δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένα τα πράγματα, τι σημαίνει δηλαδή προσθετικότητα και ποια είναι η ερμηνεία της. Τέλος, από την εμπειρία βλέπουμε ότι πολύ blending απευθύνεται τελικά σε χώρες μεσαίου εισοδήματος, ενώ ο στόχος ιδίως του Ταμείου είναι να στοχεύσει κυρίως τις εύθραυστες χώρες. Η ερώτηση λοιπόν είναι εν τέλει αυτό το blending είναι πράγματι κατάλληλο. Έχει την ικανότητα πραγματικά να φτάσει στις χώρες εκείνες οι οποίες είναι φτωχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες και δυσκολεύονται περισσότερο να ε, προμηθευτούν χρηματοδότηση. Αυτές είναι κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το EFST. Προχωρώντας, είναι σημαντικό να θυμάται κανείς και κάποιες από τις συστάσεις που έχουν γίνει για βελτίωση, γιατί Πολλής προβληματισμό έχει γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίω με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα blending και Εξωτερική συνεργασία, η οποία έχει κάνει και ορισμένε συστάσει και θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένε από αυτές. Πρώτον, η ανάγκη να χρησιμοποιηθεί περισσότερο κεφάλαιο κινήσεως, ή risk capital, εγγυήσει και επιδοτήσει επιτοκίων στο blending να βελτιωθεί, να βελτιωθεί τα συστήματα παρακολούθησης και υποβολής αναφορών, monitoring και reporting, κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα διαφανές πάντα. Και με τρόπο που να επιτρέπει και συγκρίσεις ανάμεσα στα διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται να συμμετάσχουν περισσότερο και οι επιτόπου, για παράδειγμα, αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθήσει ευρύτερη συμμετοχή μεταξύ των φορέων που προσφέρουν ε, βοήθεια. Όχι μόνο των ευρωπαϊκών, αλλά και των μη ευρωπαϊκών. Και στις χώρες εκείνες όπου θα λάβει χώρα η επένδυση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να μην συμμετάσχουν, να μην συμπεριληφθούν μονάχα στις τελευταίες φάσεις, αλλά από την αρχή, από τον σχεδιασμό της επενδύσεως για να ληφθεί υπόψη η οπτική και η προοπτική της χώρας όπου θα διεξαχθεί η επένδυση. Το βασικό καινοτόμο στοιχείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης και βασισμένο στο παραδοσιακό blending είναι η διαχείριση του κινδύνου. Αυτός είναι ένας από τους πυλώνες του προγράμματος εξωτερικών επενδύσεων. Δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ, αλλά πρόκειται για μια σημαντική καινοτομία. Και κυρίως λοιπόν το θέμα του κινδύνου. Τονίζω εδώ ένα είδος προβλήματος το οποίο αναφύεται διαρκώς, σαν, κάτι σαν εκείνο το ΚΑΤΣ 22. Ο κίνδυνος δηλαδή όταν δίνονται εγγυήσει κατά του κινδύνου να απαλλαχθεί υπερβολικά, δηλαδή να αρθούν τα κίνητρα που δίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Και τότε καταλήγουμε, μιλώντας με εμπειρογνώμονες, ότι βρίσκουν το σωστό επίπεδο του κινδύνου. Όταν όμως ρωτάτε γιατί δεν κάνετε περισσότερα για την κάλυψη του κινδύνου, Όπω εξήγησε στο παράδειγμα του κ. Σουαταρά, λένε ότι δεν θέλουν να αναταράξουν πολύ την αγορά. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε στρεβλώσει την αγορά. Αν κάνουμε περισσότερα, τότε καλύπτεται περισσότερος κίνδυνος. Και τότε υπάρχει ο κίνδυνος να σπαταλώνται τα χρήματα της ε, επένδυσης, τα δημόσια χρήματα τη επένδυση. Χρειάζεται λοιπόν η αναζήτηση μια σωστή ισορροπία που δεν είναι πάντοτε απόλυτα σαφές πώς μπορεί να γίνει. Και αυτή είναι η πρόκληση και για το EFST και από την άποψη αυτή είναι σημαντικό να εξεταστεί και η εμπειρία και κάποιων άλλων φορέων όπως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που έχει μια διευκόλυνση για τις χώρες ΑΚΕ. Υπάρχει το πλαίσιο της διευκόλυνσης, όμως όλες οι εξωτερικές διαδικασίες αναφέρονται στον κίνδυνο, αναφέρονται στην ανάλυση μεγαλύτερου κινδύνου, αλλά και λόγω της εσωτερικής λειτουργίας μπορούν εν τέλει να αναλαμβάνουν την κάλυψη μεγαλύτερων κινδύνων. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Να ολοκληρώσω λέγοντας ορισμένες, αναφερόμενες ορισμένες βασικές σκέψεις στην ανάγκη να βασιστούμε στα διδάγματα που έχουμε ήδη από τις διάφορες διευκολύνσεις ανάμειξης από, τα διάφορα, από τους διάφορους οργανισμούς αναπτυξιακής βοήθειας και βεβαίως το IFC που είναι το πιο δραστήριο για, την, ε, για τις επενδύσεις σε εύθραυστες χώρες και το θέμα της προσθετικότητας και πώς μετράται η προσθετικότητα γιατί είναι από, μια από τις βασικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι αποφάσεις για επενδύσεις. Και βεβαίως χρειάζονται και κριτήρια διαφάνειας. Και τέλος, το ζήτημα της συνοχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης με την Ευρωπαϊκή ε, Συνεργασία για την Καινοτομία. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βιλάλ, βλέπουμε ότι σημαντικές είναι και οι αρχές, αλλά σημαντικό είναι και πώς μπορούμε να εφαρμόζουμε όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Ερχόμαστε στον επόμενο μιλητή, είναι ο κύριος Χαβιέρ Σόλ από την Counter Balance, ΜΚΟ. Σε πολιτικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια ισορροπία και με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε όσα έχετε να μας πείτε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν ε, την πρόσκληση. Εγώ προέρχομαι από τη ΜΚΟ Counterbalance να μιλήσω και εξ ονόματος μιας ομάδας ε, ΜΚΟ που παρακολουθούμε την σύσταση του ε, σχεδίου εξωτερικών επενδύσεων. Ε, και αυτό γιατί έχουμε κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τους λογικούς και στόχους αυτής της επενδυτικής πρωτοβουλίας. Πρώτα απ' όλα, για την ώρα δεν είναι σαφές εάν ε, το ευρωπαϊκό επενδυτικό αυτό σχέδιο θα είναι, πραγματικά θα σημάνει την αλλαγή, γιατί είναι προσθετικότητα και προσθέμενη αξία ε, για την ανάπτυξη δεν είναι καθόλου ξεκάθαρος. Πρέπει να μάθουμε τα διδάγματα προηγούμενες ε, πρωτοβουλίες επενδυτικές, όπως έλεγε ο κύριος ε, Μπιλάλ. να δοθούν οι εγγύησεις δεν σημαίνει ότι, θα, ότι δεν θα γίνει business as usual. Δηλαδή, οι εγγύησεις δεν είναι κάτι το θαυματουργό. Αν δούμε το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, διαφορετικό επίπεδο, αλλά πολλά ελέγχθηκαν για το ΕΦΣΙ και για την προσθετικότητα. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίσης και η εντολή για εξωτερικές, ε, ε, εξωτερικό δανεισμό ακόμα και αν οι εγγυήσεις προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, σημαίνει αυτό αυτόματα ότι η τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επενδύει σε σχέδια υψηλού κινδύνου ούτε σε χώρες που θεωρούνται με υπερβολικό χρέος. Οπότε Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πραγματική προσθετικότητα για την ανάπτυξη. Τι γίνεται με την αξιολόγηση των ήδη ε, υπαρχουσών διοδοτικών δυνατοτήτων. Ε, εξεδόθη έκθεση στα τέλη του 2014 για αυτό το θέμα και εδώ περιλαμβάνονται κάποιες ε, παρατηρήσεις επικριτικού χαρακτήρα σε σχέση με τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ωστόσο, από τότε δεν έχει γίνει κάποια Αξιολόγησε από την Κομισιόν πριν την πρόταση και αυτό το επενδυτικό πλάνο. Οπότε, ποια είναι η ανάγκη για επέκταση των δανειοδοτικών μηχανισμών. Είναι ο καλύτερος τρόπος χρήσης των ευρωπαϊκών χρημάτων. Είναι κρεμή ζητήματα που δεν έχουν απαντηθεί όλα ε, ακόμη. Δεύτερο η παρατήρηση είναι ότι πιστεύουμε πως η σύνδεση με ότι έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση με την μεταναστευτική πολιτική που είναι επικίνδυνη. Εμείς θέλουμε λοιπόν να διαγραφεί αυτό το επενδυτικό σχέδιο από την βράχη πρόθεσμη πολιτική, εξωτερική πολιτική. Είναι μια κίνηση για να κινηθούν περισσότερο τα, οι θεσμοί για τα θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης και βλέπουμε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απομακρύνονται όλο ένα και περισσότερο από τους ε, στόχους αυτούς. Έχουν απομακρυνθεί και με τις πρωτοβουλίες της ε, ΕΤΕΠ και την, ε, την Υπάρχει αυτή η τάση για απομάκρυνση των τραπεζών από την ανάπτυξη και δεν θα πρέπει να είναι ο ρόλο των εθνικών αναπτυξιακών ε, τραπεζών να γίνουν οι χρηματοδότες τη Ευρώπη οχυρού. Ε, εδώ λοιπόν πρόκειται για την επέκταση μηχανισμών ανάμειξη που υποτίθεται ότι θα είναι εργαλεία αναπτυξιακά και πιστεύουμε πως αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να μείνει η αναπτυξιακή πρωτοβουλία και να μην έχει σχέση με άλλα ζητήματα. Τρίτη παρατήρηση είναι ότι αν θέλουμε αυτό το επενδυτικό σχέδιο να αποτελέσει πραγματική αναπτυξιακή ε, βοήθεια και να είναι ένα πραγματικό εργαλείο μέσο και να επιτύχει τους στόχους ε, για την επίτευξη των ε, βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Σε αυτή τη στιγμή στον κανονισμό δεν περιλαμβάνονται επαρκείς ε, κοινωνικές, περιβαλλοντικές ε, ή εργασιακές ασφαλιστικές δικλείδες, ούτε αυτές που να συνδέονται με την κοινωνική ε, πολιτική, την πολιτική για την ισότητα των φύλων. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν εγγυήσεις και μέσα στον κανονισμό να υπάρχει σταθερότερη και ξεκάθαρη γλώσσα για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των διοικητικών μηχανισμών και σε επίπεδο έργου. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί η λογοδοσία ώστε τα project τα οποία θα υποστηριχθούν να είναι ε, ξεκάθαρα για την φορολογία, να μην ευνοούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να συμβάλλουν στην ε, μόχλευση χωρίων πόρων, αλλά και θα συμβάλλουν στη ε, επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας για τις Κλιματικές Αλλαγές του Παρισιού. Τέλος, να πω ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτό το πρόγραμμα ε, ε, όπως είπα, αυτή η σύνδεση με τη μετανάστευση, τα μεταναστευτικά ζητήματα. Ταυτόχρονα όμως για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να θεωρηθεί ως ευκαιρία ώστε επιτέλους να έχει λόγο για αυτούς τους μηχανισμούς ανάμειξης που ήδη υπάρχουν σήμερα. Ιδιαίτερα δεδομένου ότι το blending αυτή η ανάμειξη παρουσιάζεται όλο ένα και περισσότερο ως ένα, ένας χάρτης, ένα προσχέδιο για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η συζήτηση για τη δημιουργία του EFSD του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για Βιώσιμης Ανάπτυξης ε, έχει να κάνει με την διαφάνεια, τη λογοδοσία. Ε, είναι μια ευκαιρία για το Κοινοβούλιο ώστε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο, ώστε να εξασφαλίσει πως αυτή η πρωτοβουλία θα είναι πραγματικά αναπτυξιακή και αυτό έχει σημασία από την πλευρά των ΜΚΟ, να εξασφαλίσουμε ότι θα στοχευθεί στην εκρίζωση της, φθο... της Ότι θα στοχεύει μάλλον στην εκρίζωση της στόχης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ε, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Uh, uh, Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ερχόμαστε στις ερωταπαντήσεις. Για τους συγκητές έχουμε δύο λεπτά για τον καθένα. Θα μιλήσουν πρώτοι η κυρία Γκάρδια Θάμπαλ από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές μας για τις παρουσιάσεις τους. Από μια πρώτη αξιολόγηση των όσων ακούσαμε και ελπίζω να συμφωνούν και οι συνάδελφοι συνεισηγητές, αν μη τι άλλο, στην ανάλυση του ΕΤΒΑ συμφωνούμε στον εντοπισμό των μεγαλύτερων προβλημάτων για την ε, πρόταση αυτή για ένα ταμείο βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι, συμφωνούμε στη διάγνωση. Ποια είναι τα προβλήματα, ποιε είναι αμφιβολίες, το ακούσαμε από τους ομιλητές μας. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που κυριαρχεί και που συζητάμε είναι πώς ε, θα βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει αυτή η προσθετικότητα με την ευρύτερη έννοια. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πλατφόρμες blending και πώς ε, μπορεί αυτή η εγκύριση να έχει μια προστιθέμενη αξία στις πλατφόρμες αυτές και προσθετικότητα υπό την έννοια ότι δεν θα χρηματοδοτήσουμε ιδιωτικά έργα που θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν θα πετάξουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις από την αγορά. Άλλα τα θέματα που μας απασχόλησαν ε, είναι ε, τι γίνεται με τη συνέχεια και τη συνέπεια των στόχων των αναπτυξιακών, αλλά όχι μόνο του συγκεκριμένου ταμείου, αλλά και άλλων προγραμμάτων που ε, εργάζονται στους ίδιους χώρους, στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές και στα ίδια θέματα. Μ' άρεσε αυτό που είπατε και πώς συνδέσατε την εκτίμηση κινδύνου με την επένδυση είναι πραγματικά κλειδί για να πιάνουν τόπο τα χρήματα. Και για τους στόχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι κάτι που μας απασχολεί και εμάς τους εισηγητές και θελήσαμε να ακούσουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα γιατί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν λίγο γενικόλογη και χρειαζόταν ε, κάποια κριτήρια πολύ πιο σαφή και συγκεκριμένα για να υπάρχει προστιθέμενη αξία και να αποφευθούν ε, επικαλύψεις με άλλα ταμεία. Ευχαριστώ και τώρα θα αφήσω το λόγο στους άλλους συναδέλφους μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους μας. Είναι πάρα πολύ σαφή και σταράτα αυτά που μας λένε και επικεντρώνονται στα πράγματα που μας ενδιαφέρουν και που συζητούμε. Υπό την έννοια αυτή ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και διαφωτιστική αυτή η συνεδρίαση. Και αυτό δεν είναι μια υποχρεωτική ε, διπλωματική πυρουέτα, το εννοώ αυτό που λέω. Ε, ίσως ε, θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Εγώ συμφωνώ με την προλαλή σας. Πολύ γενικές ερωτήσεις. Ε, αναφερθήκατε ακροθυγώς αυτές στην εισαγωγή σας, αλλά θα ήθελα λίγο να επιμείνω. Προς τον κύριο Βαταρά, μια πολύ γενική ερώτηση. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν τα πραγματικά ωφέλη για τις αφρικανικές χώρες, για την ανάπτυξή τους δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγκριθεί το σωστό εργαλείο, το χρηματοδοτικό. Και για τους κινδύνους Δύο από εσά μίλησαν για την εκτίμηση κινδύνου και την ανάλυση. Ερωτώ λοιπόν. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στη φάση εφαρμογής του Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το είπε και ο κύριος Σωταρά και η κυρία Χίφ. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο. Θα σας ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούκαν. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους ομιλητές μας για τις παρεμβάσεις τους. Είχαμε και άλλες συνεδριάσεις πρόσφατα και σήμερα μάλιστα στο Κοινοβούλιο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. και τις ε, υπηρεσίες εξωτερικής δράσης. Από τη σκοπιά της Επιτροπής Αναπτυξιακής ε, Πολιτικής θέλω να σας πω ότι ε, μας ανησυχούν οι αναφορές στο άρθρο 21 στη Συνθήκη της Λισαβόνας ή το 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλάμε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και συνεκτική πολιτική, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα φύλων, ζητήματα κλιματικών αλλαγών, φοροαποφυγής, όλα αυτά τα θέματα έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν συμπεριληφθεί. Και πρέπει να σας πω τώρα ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των συνεισηγητών. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα που πρέπει ακόμα να διευκρινιστούν. Και ισχύει και για εσάς αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που λέει ότι ωραία, έχουμε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δίνουν δάνεια και έχουμε ένα συνδυασμό χρηματοδότησης, αυτό το περίφημο blending. Όλοι αυτοί οι όμιλοι λοιπόν οι χρηματοδοτικοί που συμμετέχουν. Πώς θα υποστηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις τις υποδομές, τις κοινωνικές, στις λιγότερο επτυγμένες χώρες, σε ζώνες σειράξεων, σε ζώνες αστάθειας. Όχι μόνο στην Αφρική, αλλά και στην ανατολική μας γειτονία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ κοντά. Θυμηθείτε την κατάσταση στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και όδησηγητές τώρα. Βλέπω την κυρία Χάουταλα. Thank you Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλο το πάνελ για τις θαυμάσιες ε, παρουσιάσεις που μας επιτρέπουν να ε, καταλήξουμε και σε κάποιες τροπολογίες για την πρόταση της Κομισιόν. Ποιες συγκεκριμένες συστάσεις μπορείτε να μας δώσετε για να διασφαλιστεί η προσθετικότητα κατά για το οποίο μίλησαν λίγο πολύ όλοι οι ομιλητές και είπαν ότι θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένοι και μπορούμε να εντάξουμε στον κανονισμό κάποιες αυστηρές εγγύσεις όσον αφορά την υποχρέωση αυτών που θα τα υλοποιήσουν ότι θα σέβονται τις αρχές που επιβάλλουμε. Και για την κυρία Heath που δυστυχώ έχασε το πρώτο μέρος της παρεμβάσεω της, Παρ' όλα αυτά μιλώ για το impact investment. Θεωρείτε ότι έχει σοβαρό δυναμικό για να επιφέρει κάποια επίπτωση, impact δηλαδή στις επενδύσεις. Βλέπετε αυτό το impact investment να προωθείτε με τη νέα ρύθμιση που συζητούμε. Uh, no. Uh, Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη του πάνελ για τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Τώρα χωρισμένα σχόλια. Πρώτα, ήδη έχουμε συλλέξει εμπειρίες με το Ταμείο EFSI, για παράδειγμα. Εφόσον μια χώρα έχει καταβάλει κάποιους πόρους Το ΕΦΣΙ βάζει 5%, η χώρα μέλος βάζει 95%. Για την επένδυση, ωστόσο, η επένδυση που τελικώς υλοποιείται θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί και χωρίς χρηματοδότηση από το EFSI. Βεβαίω υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα μόχλευση. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τα επενδυτικά έργα στην Αφρική. Το λέω αυτό για να αποφύγουμε λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Δεύτερο, πώς μετρούμε την επιτυχία. Για παράδειγμα, αριθμοί θέσεων απασχολήσεως που δημιουργήθηκαν, μείωση της φτώχειας. Άλλο ερώτημα. Η Αφρική αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα δημογραφικού χαρακτήρα. Η Αφρική έχει τώρα 1,2 δισεκατομμύρια κατοίκους. Μέχρι τα τέλη, μέχρι του αιώνα θα έχει φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια. Αυτά πάντοτε σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη, το, μόνη της αυτό η Αφρική. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να γίνουν σοβαρές επενδύσεις στην παιδεία στην Αφρική. Εδώ μιλούμε ιδίως για επενδύσεις σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως η Αφρική χρειάζεται επενδύσεις στην παιδεία, ιδίως στην παιδεία των γυναικών, των νεαρών κοριτσιών, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν λες, αυτές οι προκλήσεις δημογραφικού χαρακτήρα. Χρειάζεται να αναζητηθούν λοιπόν και άλλα εργαλεία εντό εισαγωγικών για να μπορέσουν να γίνουν τέτοιε επενδύσει στην Αφρική. Τι γνώμη έχετε για αυτά, Πρόεδρο, ευχαριστώ. Νομίζω ότι ακριβώ αυτό είναι το πρόβλημα. Από τη μία μεριά Έχουμε ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τις επενδύσεις, αλλά πάντα κάνουν και μόνες τους, γιατί μπορούν να υπολογίσουν τον κίνδυνο. Από την άλλη έχουμε τις ευκαιρίες υπολογισμού του κινδύνου, αλλά και ευκαιρίες για δάνεια. Πόσο όμως είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε τον κίνδυνο, να χάσουμε πόρους από τον προπολογισμό που θα διαθέσουν σε τις επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρκα. Εσείς κύριε Χάουσερ τώρα. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Μία σύντομη ερώτηση για την κυρία Χίθ, η οποία εξήγησε κυρίως έργα κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα και πώς αξιολογούνται αυτά. Πώς μπορεί το Ταμείο EFSD να φροντίσει να αποφευθούν ανισότητες και ποιους κινδύνους βλέπετε, ποιες επενδύσεις βλέπετε να φέρουν τον κίνδυνο ενίσχυση τελικά της ανισότητας. Άλλος ε, κανείς δεν βλέπω άλλα μέλη να ζητούν το λόγο. Επιστρέφω το μικρόφωνο στο πάνελ. Ποιος επιθυμεί να απαντήσει. Ο Αταρά. Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την επίπτωση που μπορούσε να έχει ε, στην ανάπτυξη ε, της Αφρικής ε, το σωστό ταμείο. Ο αντίκτυπος είναι πολλαπλός. Πρώτο στοιχείο η αυτονομία. Ο ιδιωτικός τομέας στην Αφρική δεν ζητάει χρηματοδότηση για τη χρηματοδότηση. Η αυτονομία ζητάει ανεξαρτησία. Γίνεται λόγος για επιδοτήσεις, αλλά σήμερα οι επιδοτήσεις, οι κρατικές ενισχύσεις δεν είναι αυτό που ζητούν οι εταιρείε θέλουν δάνεια, αλλά να είναι σε θέση να τα αποπληρώνουν. Ε, υπάρχει μια μόχλευση και πρέπει να δράξουν την ευκαιρία. Οι κρατικές ενισχύσεις δεν πρέπει να πηγαίνουν για ε, τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά για το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό που ζητούν οι επιχειρήσεις είναι αυτόνομη. Το δεύτερο είναι η αντοχή και η αθεκτικότητα ε, στις παγκόσμιες αγορές. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές οι αφρικανικέ εταιρείε. Υπάρχουν προβλήματα προτύπων, προδιαγραφών, time to market, δηλαδή έγκαιρη διάθεση στην αγορά των προϊόντων. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε εταιρείε από την Ασία, Φερρυπίν. Αυτό είναι ένα από τα ωφέλη. Μετά η ποιότητα ζωή. το επίπεδο διαβίωση. Δηλαδή είναι άλλο να εργάζεται, ο άλλο να ε, μπορεί να έχει ένα στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης και εδώ θα αφαιρθώ λίγο στη μετανάστευση γιατί γίνεται μέγας λόγος για τη μετανάστευση. Δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα εκεί, είναι σημαντικό να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και να πούμε ποια είναι η ευθύνη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το έχω ζήσει και εγώ ε, ως μετανάστης εντός αγωγικών. Εγώ στην Αφρική μεγάλωσα. Στην Αφρική όταν είναι νέος τι σου λέει η τηλεόραση, η διαφήμιση, τα μίντια. Ένα όνειρο σου παρουσιάζουν. Η Ευρώπη, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ονειρεμένοι τόποι. Δεν ε, σου δείχνουν την πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχει ευθύνη των ε, ντόπιων αρχών για το τι δείχνουν τα μίντια. Θα μπορούσε ε, η τηλεόραση να δείχνει εκπομπές για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, για την επιχειρηματικότητα. Έρχεται ο νέος κομμένος από την οικογένειά του, βρίσκεται στην Ευρώπη ε, τελείως ε, αβοήθητος και ανήμπορος. Ε, δηλαδή θα πρέπει και οι ντόπιοι πολιτικοί να ευαισθητοποιηθούν και να παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα. Μετά έγινε μια ερώτηση για το θετικό αντίκτυπο. Πώς μπορεί δηλαδή να επηρεάσει ένα τέτοιο πρόγραμμα θετικά την οικονομία και την ανάπτυξη έχει σημασία να εμπλακούν και κάποιοι τρίτοι ε, ε, παίκτες εκεί. Δηλαδή, ε, όχι κατά ανάγκη οι ντόπιε τράπεζες και οι ντόπιοι πολιτικοί, κάποιοι μεσολαβητές, κάποιες εταιρείες συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, λογιστών που κάνουν το business plan της επιχείρησης, που έχουν την καλύτερη γνώση των πραγμάτων, Πολλές φορές έχουμε επιχειρήσει με διπλά βιβλία. Έχουν άλλα βιβλία για την εφορία της χώρας και άλλα βιβλία για τον επενδυτή. Ε, θα πρέπει κάθε φορά να ξέρουμε ποια είναι τα σωστά στοιχεία και ποια τα αξιόπιστα. Και πώς θα ε, βγει από αυτή την κρίση η Αφρική με την παιδεία βεβαίως την εκπαίδευση και για την επιχειρηματικότητα. Βλέπετε σήμερα τι συμβαίνει οι οικογένειε στην Αφρική δεν έχουν πάντα αυτό το αντανακλαστικό ε, της αποταμιεύση, τη προώθηση των νέων. Είναι και αυτό το, κάτι το οποίο διδάσκεται το επιχείρημα για να αλλάξει η νοοτροπία και η κουλτούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάνει προτάσεις για την επιχειρηματικότητα των μεταναστών, για να χειραφετηθούν και να ενδυναμωθούν περισσότερο οι μετανάστες. Μπορεί να είναι ένα μικρό τμήμα και αυτό της λύσης. Πάντως θα πρέπει εμείς να ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Η κυρία Χίθ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις ομαδικά. Εμείς αναζητούμε όχι μόνο την υγεία μιας συμμεμονωμένης εταιρεία, αλλά μιας ολόκληρης οικονομίας. Και θέλω να δώσω μια παρομοίωση και ζητώ συγγνώμη που είμαι κάπως απλοϊκή, αλλά εάν επενδύσεις σε μια εταιρεία που ρηπαίνει ένα ποτάμι, οι εταιρείε που, είναι, που υπάρχουν πιο κάτω στο ποτάμι ε, θα ζημιωθούν από αυτό. Γι' αυτό και θα πρέπει ε, να προσέχουμε συνολικά το τι επενδύσεις προωθούμε και θέλω να τονίσω την ανάγκη να εξετάσουμε όλη την εργασία δέουσας επιμέλειες που έχει γίνει από την ε, επενδυτική ε, κοινότητα. Επίσης θέλω να πω ότι ο βασικός ρόλος των βιώσιμων στόχων ανάπτυξη, ανάπτυξης ε, είναι σωστό να στοχεύσουν επενδύσεις όχι μόνο για την εξασφάλιση αλλά και για την ε, στόχευση σε σωστές, σωστού είδους επενδύσεις. Τώρα, επενδύσεις και αντίκτυπος αυτών. Θα έλεγα ότι κάθε επένδυση έχει αντίκτυπο. Εμείς μετράμε όμως μόνο το θετικό και αντίκτυπο και αυτόν συζητάμε. Όμως όλες οι επενδύσεις έχουν ένα κάποιο αντίκτυπο. Όταν προσπαθούμε να μετρήσουμε την βιώσιμο αντίκτυπο μια τέτοια επένδυση, θα θέλαμε να μετρήσουμε και το πόσο βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται, ε, αλλά ακόμα δεν έχουμε τον τρόπο να το μετρήσουμε. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια και την, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Επίσης, οι κοινωνικο-οικονομικά projects και πράγματα που μειώνουν την ανισότητα. Δεν είμαι σε θέση να πω ποιο είδους επενδύσεις είναι οι πιο επικίνδυνες, όμως θέλω να επαναλάβω ότι αυτό που βλέπουμε επανειλημμένα είναι ότι η ποιότητα των θέσεων που δημιουργούνται και η σχέση ανάμεσα στην εταιρεία και τους εργαζόμενούς της είναι πολύ σημαντικό κριτήριο για να αξιολογήσουμε κατά πόσο αυτή η εταιρεία ε, προωθεί την ισότητα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπιλάλε, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι ο κίνδυνος, οι επικίνδυνες επενδύσεις είναι πραγματικό εμπόδιο για τον ιδιωτικό τομέα. Αν μιλάμε για ιδιωτικές επενδύσεις ε, στην Αφρική αλλά και στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν επενδύουν ιδιώτες. Ε, είτε επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, είτε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λένε γιατί δεν γίνεται η επένδυση. Άρα Πολλές φορές, πολλές φορές όμως οι ιδιαίτερες αντιλαμβάνονται το κίνδυνο πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό γίνεται και η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε πρώτα αυτό το θέμα, ότι ορισμένες ε, επενδύσεις είναι όντως πιο επικίνδυνες, ιδιαίτερα στα ευάλωτα κράτη. Έχουμε διαφόρων ειδών κινδύνους, ε, ε, το νόμισμα, πολιτική κίνδυνη, και υπάρχει και αυτό η διαφορά αντίληψης για το κάθε είδους κινδύνου. Είναι σημαντικό λοιπόν να σημάνει ε, τη διαφορά αυτό το σχέδιο, το επενδυτικό, όσον αφορά τις ρηψοκίνδυνες ε, επενδύσεις. Επίση αναφέρθηκε ότι υπάρχει περισσότερη ανάγκη ε, συνοδείας τεχνικής αρρωγής και αυτό μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο του σχεδίου του επενδυτικού. Για να λειτουργήσουν όλα αυτά χρειάζεται να ισχύσουν διάφορες αρχές που θα κατευθύνουν και θα εξασφαλίζουν τις αρχές, αλλά επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και τις διαδικασίες, πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να χτίσουμε στο τι κάνουν, πάνω σε αυτό που μάλλον ε, ε, κάνουν οι ε, θεσμικοί επενδυτές και η θεσμική χρηματοδότηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Και επίση να μην κάνουμε υπερβολικά πολλά εφόσον ισχύουν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι, να μην βάλουμε πολλούς όρους, γιατί αν απαιτήσουμε και αντίκτυπο ε, αναπτυξιακό για τους επενδυτέ. Ε, δεν θα βρούμε αρκετού επενδυτέ, γιατί θα είναι πολύ δύσκολη η τήρηση όλων των κριτηρίων και των όρων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλ, τελευταίος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός. Yes, I will... Ναι, θα επανέλθω σε μερικά από όσα με ρωτήσατε. Πρώτον, το πιο δύσκολο είναι η προσθετικότητα. Πώς θα ε, ορίζονται ε, τα έργα υψηλού κινδύνου. Δεν είναι μόνο οικονομικά τα κριτήρια, αλλά είναι και το θέμα της προσθετικότητας. Είναι οι λεγόμενες ΣΔΙΤ, συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και άλλα κριτήρια που πρέπει να μελετήσουμε. Ε, περιβαλλοντικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια, ανισότητες, όλα αυτά συνυπολογίζονται ε, στους δείκτες που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθούν και να εκτιμηθούν ε, τα προγράμματα και τα έργα ανάλογα με το ρίσκο. Τα ίδια ισχύουν και με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Υπάρχει ένα βαθμολόγιο δικτών ε, που δημιουργήθηκε, τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται πάντα το χ, αλλά είναι αντίστοιχο το σύστημα όπου μπορούν να κάνουν προτάσεις οι διάφοροι ενεχόμενοι και ενδιαφερόμενοι για να δημιουργηθούν οι σωστοί δείκτες που θα μετρούν το ρίσκο κάθε φορά της επένδυσης. Δεν είναι μόνο οικονομική όρη. Μετά, ασφαλιστικές δικλείδες, τι μπορεί να γίνει συγκεκριμένα Υπάρχουν διάφορες ιδέες για να σας δώσω μερικά παραδείγματα για την κλιματική αλλαγή. Αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά καινοτόμα έργα για την πιο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των ε, χωρών εταίρων, δεν υπάρχει χώρος ε, για έργα, ας πούμε, σε ορυκτά καύσιμα. Ας πούμε, ε, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, κάποια έργα ε, που είναι σε συγκεκριμένες χώρες που δεν συνεργάζονται, επίσης δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Έκθεση αναχώρα, ε, πεπραγμένων και δραστηριοτήτων είναι κάτι που απαιτείται. Ορίστε μερικά παραδείγματα και επίσης θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποιους ορισμούς. Οι αναπτυξιακές τράπεζες, τα επενδυτικά ιδρύματα, τα χρηματοπιστωτικά έχουν το ρόλο τους, αλλά έχει διακριτό ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι κανένα από τα έργα που χρηματοδοτούνται δεν παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να είναι αποκλειστικότητα, η εκτίμηση δηλαδή της κάθε τράπεζας, αλλά και της Κομισιόν. Α, μάλιστα, ακριβώς τώρα ερχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα λεπτό, το πολύ δύο, άντε. Παρακαλώ, Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, ποιος θα πάρει το λόγο. Τμήματάρχης για τα χρηματοδοτικά μέσα και αρμόδιος για το ε, σχεδιασμό των επενδύσεων. Άκουσα πολύ προσεκτικά και προσπάθησα να βρω ένα θέμα στο οποίο να διαφωνώ και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Και εμείς την ίδια ανάλυση έχουμε και ε, ο προγραμματισμός για τις εξωτερικές επενδύσεις είναι κάτι που θέλουμε και εμείς για να επιταχυνθούν τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα και να υπάρξει το blending. Δύο σχόλια. Για την εκπαίδευση και την παιδεία χρειάζεται προσοχή εδώ πιστεύω. Να μην ε, διαφημίζουμε το blending ως πανάκια για όλα τα δεινά του κόσμου. Αυτό το blending απευθύνεται σε συγκεκριμένα έργα. Υπάρχουν ε, έργα και έργα. Μερικά χρηματοδοτούνται από δάνεια και άλλα από ε, κρατικές ενισχύσεις ή από ε, χρηματοδότηση που δεν επιστρέφεται. Επίσης, υπάρχει εντύπωση ότι γίνεται μια συναλλαγή ανάμεσα και με ανταλλάγματα σε διάφορους στόχους. Όταν θέλει κάποιος να έχει μεγάλη προσθετικότητα, ε, είναι πολύ διαφορετικές οι χώρες μεταξύ τους, οι λιγότερο αναπτυσσμένες χώρες. Και δεν μπορούμε ταυτόχρονα να έχουμε ε, όλα τα κριτήρια και όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες που αναφέρατε. Στην πράξη τι βλέπουμε. Ας πούμε για τα μέσα για τις μικρομεσαίες που αναφερθήκατε προηγουμένως. Ο, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πας στη μεγαλύτερη τράπεζα, ε, στην Ιγυρία ας πούμε, μια πιο ανεπτυγμένη χώρα, γιατί είναι πιο εύκολο για τις τράπεζες αυτές να χρηματοδοτήσουν το εν έργο ε, να, και να ελέγξουν αν πληρούνται τα κριτήρια. Και είναι πιο δύσκολο να πας σε μια πιο μικρή ε, τράπεζα, σε ένα ίδρυμα που έχει διαμεσολαβητικό ρόλο, που δεν σε γνωρίζει, που δεν ξέρει την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορούν όλοι οι στόχοι να πληρούνται ταυτόχρονα. Κατά τα άλλα συμφωνώ με τις παρουσιάσεις. Ευχαριστώ. Okay, thank you so much. Uh, next one is DG. Ευχαριστώ. DG Near, κύριε Μάρτινς. Ε, ε, ε ευχαριστώ. Πληματάρχης σχεδιασμού. Και υπεύθυνο της Γενικής μου Διεύθυνσης για σχεδιασμού επενδύσεων. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε τις απόψεις του πάνελ, γιατί έχουμε και πολύ διαφορετικές απόψεις σε ό,τι αφορά το, τον σχεδιασμό εξωτερικών επενδύσεων. Όμως, οι ανησυχίες μας είναι ίδιες, όπως προσθετικότητα, λογοδοσία, διαφάνεια. Αυτές τις ανησυχίες τις μοιραζόμαστε και εμείς από τότε που αρχίσαμε πέρσι να κάνουμε το σχεδιασμό και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διαδικασίες και να έχουμε και συνέχεια και των μελλοντικών έργων του, ε, του σχεδιασμού με τον ίδιο τρόπο που έχουμε κάνει ως τώρα. Δεν αρχίζουμε δηλαδή από το μηδέν. Αρχίζουμε από μια στέρεα βάση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχουμε φτάσει εκεί που είμαστε σήμερα, προσπαθούμε να κάνουμε ένα άλμα από αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα σε μια νέα κατάσταση για τον εξωτερικό επενδυτικό σχεδιασμό που να μπορέσει να αντιμετωπίσει καλύτερα τις ε, προκλήσεις και όπως είπε ο συνάδελφός μου προηγουμένως βεβαίως πρόκειται για ένα μέσον, ένα μηχανισμό που έχει κάποια όρια. Είναι σημαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι ο μηχανισμός αυτός, το blending δηλαδή στην εξωτερική συνεργασία και οι εγγύησει που σχεδιάζουμε είναι ένα μικρό μόνο μέρος του συνόλου των χρηματοδοτήσεων. Μιλούμε δηλαδή για 10 έως 12% των συνολικών χρηματοδοτήσεων διότι παραπάνω από 80% εξακολουθούν να είναι επιχορηγήσεις, grants και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη για να μην χάσουμε την οπτική, την, την, τις σωστές διαστάσεις. Και για να ξέρουμε και το blending τέλο πάντων τι δυνατότητες έχει να επηρεάσει τον πραγματικό κόσμο. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μαζί και με τους προλαλήσατε συναδέλφους μου, λέγω κι εγώ ότι μου φάνηκε πολύ χρήσιμη η συζήτηση και η συμμετοχή των μελών του πάνελ για να αντιληφθούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ένα καινοτόμο σύστημα όπως αυτό που σχεδιάζουμε τώρα. Με ενδιαφέρει επίσης η συνέχεια της, η συνοχή καλύτερα της πολιτικής για την ανάπτυξη νέα πρωτοβουλία μέσα στα πλαίσια του θεματολογίου της μετανάστευσης και των πορισμάτων του περασμένου Ιουνίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το ζήτημα είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και επομένως οι ρίζες της μετανάστευσης. Επισημένω στους αξιότιμους βουλευτές ότι οι χρηματοδοτικές πηγές, EDF, DCI, έχουν δικές τους απαιτήσεις, στόχους, νομική βάση όσον αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης, τα κριτήρια παροχής βοήθειας και ούτω καθεξής. Σίγουρα αυτό θα ληφθεί υπόψη, είμαι βέβαιος. Δεύτερο, και όσον αφορά την χρήση του External Investment Plan, θα εξετάσει τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις για δημιουργία απασχόλησης και όχι τις πολύ βραχυπρόθεσμες που αντιμετωπίζονται για παράδειγμα με άλλους τρόπους όπως το Trust Fund για την αντιμετώπιση επίγουσών περιστάσεων. Για την προσθετικότητα θεωρώ ότι είναι σημαντικό το πραγματικό τεστ, η πραγματική δοκιμασία για το μηχανισμό θα είναι η διοχέτευση ιδιωτικών πόρων και δημοσίων επενδύσεων σε εύθραστες χώρες, θεωρώ ότι για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η χρηστή διοίκηση, με το πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις από τα συμβούλια για, τις, ε, την δομή των επενδύσεων, καθώς επίσης και τους ε, κινδύνους μεταξύ αυτών και τους πολιτικούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ τα μέλη του πάνελ, τα οποία μας δίδαξαν πολλά από την εμπειρία τους. Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να τα περιλάβουμε όλα αυτά στην νομοθετική μας πρόταση. Νομίζω να συνεχίσουμε αμέσως, διότι δεν μας μένει περισσότερο από μία ώρα. Να είμαστε λοιπόν όσο γίνεται πιο αποδοτικοί θα παρακαλέσω τον κύριο Μπέρντ, τον κύριο Αντρέασεν, τον κύριο Τζόνς και τον κύριο Παολούτσι να έλθουν εδώ στα έδρανα του Προεδρείου για να προχωρήσουμε. Όπως ξέρετε, βασική δραστηριότητα του Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να δίνει δάνεια και αν αυτά πάνε τελικά στην κατανάλωση είναι καλή η απόδοση των επενδύσεων αλλά δεν είναι αυτά που θέλουν να δουν οι δανειοδότες. Η πρωτοβουλία δημιουργίας του Ταμείου αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια ευκαιρία να δραστηριοποιηθούμε και να προχωρήσουμε με το σωστό τρόπο. Να δώσω λοιπόν αμέσως τον λόγο στον κύριο Μάρκους Μπέαντ, που είναι τμήματάρχης επιχειρηματική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της EIB, η οποία λαμβάνει την ευκαιρία για να αναλάβει χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Δεν είναι εύκολο το έργο της, γιατί από την άλλη μεριά έχουμε και την περίφημη Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, έχουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχουμε διάφορους θεσμούς οι οποίοι παρακολουθούν πολύ προσεκτικά το τι συμβαίνει. Ελπίζω ποτέ να μην χρειαστούμε για τις δραστηριότητε αυτές να εμπλέξουμε και την όλη αυτή την υπηρεσία καταπολέμησης απατών. Και ε, ε, τέλει, για να μην μακρηγορώ, να δώσω το λόγο στον κύριο Μπέντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μοιραστούμε μαζί σας τις απόψεις μας με το Κοινοβούλιο. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλωσορίζει την πρόταση αυτή για το Ταμείο ε, Βιώσιμης Ανάπτυξης. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι ακόμα τα προβλήματα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και να εργαστούμε όσο γίνεται περισσότερο με εταίρους εξωτερικούς, όπως ε, είναι ε, άλλες τράπεζες. Εμείς είμαστε η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, έχουμε το ένα νέο ταμείο και το τμήμα των εγγύσεων. Σύμφωνα με τη συνθήκη, έχουμε συγκεκριμένους στόχους και ρόλους. Να υποστηρίξουμε όχι την πολιτική τόσο πολύ, στη ε, συμπροματικότητα με εφιστάμενα ε, χρηματοδοτικά μέσα, ε, από την τραπεζική σκοπιά, να δώσουμε μια τραπεζική διάσταση στο Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Δεύτερον, μπορούμε να συνεισφέρουμε στην τεχνική παρακολούθηση του νέου ε, εργαλείου, γιατί είναι ένα τραπεζικό σύστημα, ένα σύστημα εγγυήσεων, αλλά εγγύσεις και τα δάνεια διαφέρουν πάρα πολύ από τις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, τα grants. Ε, και επίσης ε, αυτό είναι ένα κίνδυνος για τον προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια επιπλέον ε, των προβλέψεων ε, καλύπτονται και προστατεύονται. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το χαμηλότερο αντίκτυπο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στη συνέχεια, μαζί με τα υφιστάμενα μέσα που ήδη υλοποιούμε ως τράπεζα, ACPIF ε, για τις χώρες ΑΚΕ που αναφέρθηκε προηγουμένως, το επενδυτικό ταμείο για χώρες ΑΚΕ, χρησιμοποιούμε τις εγγυήσεις για τα δάνεια και θα ήθελα να αναφέρω σε συντομία τα εξή ε, σημαντικά για μας θέματα. Πρώτον, θα πρέπει να αποφύγουμε επικαλύψεις με υφιστάμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα ή μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι εταίροι μας, είτε αυτά είναι διμερεί είτε είναι πολυμερή χρηματοδοτικά μέσα και ιδρύματα. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μακροπροσθετικότητα. Αλλά και η μικροπροσθετικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως ακούσαμε στο προηγούμενο πάνελ. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε ε, ένα σύστημα πάρα πολύ συνεκτικό και αυστηρό για τη ε, μέτρηση του αντικτύπου, έτσι ώστε ε, να έχουμε το, την απήχηση που επιδιώκουμε κάθε φορά ε, με τα συγκεκριμένα στάνταρ και προδιαγραφές. Αυτό το λέει και το βαθμολόγιο του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων που αναφέρθηκε προηγουμένως του ΕΦΣΥ που βασίστηκε στο ίδιο πλαίσιο της ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Επόμενο θέμα σημαντικό για μας ε, είναι να είναι δεδομένη η τεχνική αρτιότητα ε, των θεμάτων, ε, των προγραμμάτων αυτών, να μην έχουμε σπατάλη χρημάτων και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα, είναι περίπλοκο το Ταμείο και εμείς με χαρά να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με βάση την ε, εμπειρία που έχουμε όλο αυτό των ετών, όχι μόνο ως τράπεζα, αλλά και ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξέρουμε ε, τις προδιαγραφές, τα πρότυπα και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άλλο επίσης σημαντικό θέμα κατά την άποψή μας είναι να υπάρχει μια σωστή ε, δομή διακυβέρνησης του Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης συνολικά και της διευκόλυνσης εγγύησεων, διότι ουσιαστικά ε, συνεργαζόμαστε και με θεσμικά ιδρύματα και όργανα εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι καλό να συνεργάζεσαι με του δικού σου, με τη δική σου οικογένεια, α πούμε, αλλά έχουμε και διμερεί και πολυμερεί σχέσει με ιδρύματα εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ιδιωτικό τομέα. Εξάλλου, γι' αυτό έχει σχεδιαστεί το ίδιο το μέσο. Θα πρέπει να υπάρχει χρηστή διακυβέρνηση και ταυτόχρονα να αποφεύγουμε επικαλύψει. Ε, για διάφορα συστήματα που υπάρχουν και πρωτοβολίες ε, ε, στην Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε ήδη μια εντολή για εξωτερική ε, δανειοδότηση και δεν χρειάζεται να στήσουμε νέες δομές στο Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μπορούν να συνεργαστούν με τις δικές μας υφιστάμενες δομές. Για να ολοκληρώνω, στα πλαίσια όλων αυτών, Η πρόταση του Συμβουλίου που καταρτίστηκε τα τέλη του 2016 απαντά σε πολλά από τα ζητήματα αυτά και βασίζεται σε μια συναντήληψη που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνδιαχείριση ενδεχομένω ή πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς τη διαχείριση της ευκόλης εγγύσεων έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αξιοποίηση της ε, πραγματογνωμοσύνης και της εμπειρογνωμοσύνης που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όσο γίνεται περισσότερα αποτελέσματα και μεγαλύτερο αντίκτυπο. Στο Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξη και προστατεύοντα πάντα τον ευρωπαϊκό προπολογισμό από του διαφορού κινδύνου. Μέχρι στιγμής είναι εξαιρετική η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο προηγούμενο πάνελ έτσι δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα. Πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στον κίνδυνο και την απόδοση. Αναφέρθηκε ένα διαφορετικό μέσο, το ELM, που έχει ένα πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστή και είναι διαφορετικό ως προς την εστίαση του από το δικό μας, ε, το νέο ταμείο. Θα πρέπει το Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες και στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε ήδη κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο ε, να στήσουμε ένα σύστημα συνεργασίας με τους εταίρους μας, ιδιαίτερα σε διμερές επίπεδο, αλλά και σε πολυμερές επίπεδο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, έχουμε διπλό ρόλο ως ευρωπαϊκό όργανο από τη μια και από την άλλη ως ένας μεγάλος επενδυτικός ε, όμιλος σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ ε, Μάρκους Πέρντ. Ερχόμαι στον επόμενο που είναι ο κύριος Αντριάσεν, Γενικός Διευθυντής του EDFI. Πολύ ευχαριστώ έχουμε κοντά μας. Σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε ποιος είναι ο στόχος του δικού σας οργανισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε ε, μαζί με τους άλλους συναδελφούς μου εδώ. Ε, θα αναφερθώ σε δύο βασικά θέματα. Πρώτο, γιατί είναι σωστό να επεκταθεί η χρηματοδότηση για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξή του και θα έρθω και σε ορισμένα που κάνουν οι ε, χρηματοδοτικοί οργανισμοί. Πρώτα, η επέκταση χρηματοδότησης για ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Ίσως να είναι προφανές, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να τονιστεί επαρκώς. Ότι δηλαδή η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμη για την με συλλογική προσπάθεια επιτυχία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του 2030 και ιδίω για τους στόχους μείωσης της φτώχειας, δημιουργίας απασχόλησης και ε, αντιμετώπισης της ε, κλιματικής αλλαγής. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι έχει πέσει κάτω από το 10% για πρώτη φορά στην ιστορία το παγκόσμιο επίπεδο φτώχειας και μεγάλη πρόοδος που έχει γίνει ιδίως τις τελευταίες δύο τρεις δεκαετίες ήταν το αποτέλεσμα συνδυασμού βελτιωμένων πολιτικών αλλά και ενός μοντέλου ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Και το EFSD που δίνει ιδιαίτερο φως ε, στον ιδιωτικό τομέα προσπαθεί αυτό ακριβώς να επιτύχει και βλέπουμε ε, με την πάροδο των ετών ότι η απασχόληση είναι το βασικό κανάλι μέσω από το οποίο βγαίνουν οι φτωχοί από τη φτώχεια και μέσα από την προσπάθεια αυτή 9 στις 10 δουλειές σε αναπτυσσόμενες χώρες δημιουργούνται και διατηρούνται. Χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο τους σπάνιους δημόσιους πόρους, να καλύψουμε μεγάλα δημοσιονομικά επενδυτικά κενά σε χώρες όπως αυτές που αναφέρθηκε, αναφέρθηκε προηγουμένως συναδελφή μου ως low DFI countries. Λίγα τώρα για την εντολή που έχουν οι οργανισμοί του ομίλου μας. Εμείς επενδύουμε το ίδιο όπως και οι συνάδελφοί μας σε άλλα ε, θεσμικά όργανα για να βελτιώσουμε την απασχόληση και να μειώσουμε τη φτώχεια. Ε, τα όσα έχουμε επιτύχει τα τελευταία δέκα χρόνια δείχνουν ότι οι δημόσιοι πόροι μπορούν να στηρίξουν επιχειρήσεις και στον ιδιωτικό τομέα για να επιτύχουν ανάπτυξη και το επιχειρήν είναι το κλειδί για τη δημιουργία της βιώσιμης ανάπτυξης. Πιστεύουμε ακόμη ότι ως χρηματοδοτικοί οργανισμοί πρέπει να δείχνουμε τον δρόμο και τις τάσεις, να διαμορφώνουμε τις τάσεις δηλαδή στις αγορές όπου οι επενδυτές ακόμη δεν τολμούν να επενδύσουν. Λίγα λόγια για τον ομιλό μας, 15 ε, επενδυτικών χρηματοδοτικών ε, ιδρυμάτων Έχουμε σημειώσει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Έχουμε τριπλασιάσει τις, ε, ε, το, τον επενδυτικό μας όγκο, ιδίως σε χώρες της ε, υποσαχάριας Αφρικής, όπου οδεύει το 1 τρίτο περίπου των επενδύσεών μας, ιδίως σε έργα υποδομής και κυρίως για καθαρή ενέργεια και για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Συλλογικά υποστηρίζουμε εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στις χώρες αυτές και υποστηρίζουμε και αιτήσεις πληρωμές δισεκατομμυρίων ευρώ για καταβολή φόρων. Πιστεύουμε ότι οι στρατηγικές όπως του EFSD μπορούν να βοηθήσουν να επιταχυνθεί η προσπάθεια για να φτάσουμε τους παγκόσμιους στόχους ε, ανάπτυξης και έχουμε πολύ θετικές εμπειρίες σε συνεργασία με τους ε, θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε μια πρωτοβουλία που επιγράφεται ηλεκτροδότηση και εκεί ε, κάνουμε επενδύσεις για να επιταχύνουμε την ηλεκτροδότηση σε φτωχές χώρες και φτωχές περιοχές. Σχέδια του EFSD, τα σχέδια τα οποία εμείς στον όμιλό μας ασφαλώς καλωσορίζουμε και αναμένουμε να εμπλακούμε με, τα χρηματοδοτικό, με τους χρηματοδοτικούς μας μηχανισμούς όταν θα είναι έτοιμο, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη προγραμμάτων μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού αυτού, για την επέκταση επενδύσεων σε χώρες έφραυτες και όπου σημειώνονται συγκρούσεις, να ενισχύσουμε τοπική χρηματοδότηση, εκεί όπου αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αρκετά όσο θα θέλαμε δηλαδή στις περιοχές αυτές με τους δικούς μας πόρους και από μόνοι μας και γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεργασίες με μηχανισμούς όπως το EFST, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με ανάπτυξη αγορών, αυτό έχει σχέση με ανάπτυξη αγορών, αλλά και βέβαια και με τους σημαντικούς κινδύνους των αγορών αυτών. Και κάποια από τα θεσμικά κολλήματα που αντιμετωπίζουμε ε, σημαίνουν ότι δεν μπορούμε να διοχετεύσουμε πολύ σημαντικούς πόρους προς αυτές τις αγορές. Θέλουμε επίσης οι ιδιοκτήτες μας εντός εισαγωγικών, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που βάζουν πολιτικές προτεραιότητες και μας προσφέρουν τις αναγκαίες ε, ε, ε, δεξιότητες. Πέντε, πέντε κύρια σημεία τώρα σε σχέση με, τα, με το σχεδιασμό του EFSD. Πρώτον, πιστεύουμε ότι αποτελεί ορθή χρήση των πόρων να υπάρχει δηλαδή εγγύηση χρηματοδότησης όπως αυτή που προτείνεται σε γενικούς όρους και που μπορεί να βοηθήσει στην στήριξη της ανάπτυξης σε χώρες κλειδιά χωρίς να μειώσει σημαντικά τους χρηματοδοτικούς πόρους με τρόπο τεχνικά ορθό. Δεύτερο, μας φαίνονται σωστά σωστή η ικανότητα του σχεδίου να χρησιμοποιήσει ποικιλία χρηματοδοτικών οργανισμών όπως εξηγήθηκε προηγουμένως ένα μέρος μόνο των ευρωπαϊκών blending instruments έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, μόνο ένα 5%. Με το νέο σχεδιασμό υπάρχει μεγάλη δυνατότητα επέκτασης για να συμμετάσχουν και οργανισμοί όπως ο δικός μας που έχουμε εμπειρία από συνεργασία με χώρες όπως αυτές που αποτελούν τώρα τις χώρες στόχους και σε μικρής κλίμακας έργα και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο και να διοχετεύσουμε χρήματα και σε έργα του ιδιωτικού τομέα. Τρίτο, η ανάγκη ισχυρής διακυβέρνησης και διαφάνειας όταν ε, διατίθεται δηλαδή δημόσια και ιδιωτικά χρήματα σε δύο Έχουμε τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρίας σε χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Πολλά από τα διδάγματά μας τα λάβαμε από τη χρηματοδότηση και ευρωπαϊκών χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζουμε ότι επί του παρόντος υπάρχει ανάγκη να ενισχυθούν τα μέτρα του blended financing, του, της ανάμεικτης χρηματοδότησης δηλαδή, χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των, της ανάμεικτης χρηματοδότησης για να στοχευτεί ο ιδιωτικός τομέας. Να παρακολουθείτε η αγορά προσεκτικά και να συνδυαστούν και με τι χρηματοδοτήσει του Ταμείου πράσινη ανάπτυξη. Και για τη χρήση τη ανάμετρης χρηματοδότηση σε επιχειρήσει του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε προσκαλέσει και άλλου χρηματοδοτικού οργανισμού να υποβάλουν ε, σχετικέ κατευθυντήριες γραμμέ. και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον για τι κυβερνήσει να ακολουθήσουν παρόμοιο δρόμο. Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε και έρχομαι στην προσθετικότητα ότι αν θέλουμε οι μηχανισμοί αυτοί να έχουν προσθετικό χαρακτήρα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και πιο ρηψοκίνδυνες επενδύσεις από αυτές που χρηματοδοτούν τώρα οι θεσμοί. Και ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό θα είναι να ρηχθεί το βάρος σε μια προσπάθεια να προωθούνται ε, σωστές προτάσεις. και να διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται υπερβολική χρηματοδότηση ορισμένων στόχων. Πολλοί μιλούν για υψηλά πρότυπα. Υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικά και διακυβέρνησης είναι απολύτως σημαντικά, ιδίως όταν επενδύεται σε αγορές που δεν διέπονται από νομοθεσία ικανή να κατευθύνει ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι έχουν αναλάβει ρόλο προτύπου για τα πρότυπα οι οργανισμοί μας είναι ε, ήδη ρυθμισμένοι. Τέλος, και αυτό εφαρμόζεται και για τους ε, εναρμονισμένους δείκτες αντικτύπου. Χαίρομαι επίσης για το γεγονό ότι οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί του EFST στηρίζονται και σε σχέδια για ε, παροχή τεχνικής βοήθειας, διότι η απλή χρηματοδότηση έργων δεν αρκεί για να φτάσουμε στους στόχους που έχουμε για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και είναι καλό που βλέπω ότι υπάρχει ένα συνολικό πακέτο προσεγγίσεων και μέτρων. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τον επικεφαλής του Γραφείου Βρυξελών τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. τον κύριο Μασιμιλιάνο Παολούτσι, λέει ο πρόεδρος. Τι έκανα, βιάστηκα. Όχι. Ας πάμε λοιπόν με τη σειρά. Είναι ο κύριος Γκίλιν Jones, που είναι επικεφαλής του, του Γραφείου των Βρυξελών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της περίφημης BERD. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσουμε για αυτό το πρόγραμμα ΕΤΒΑ. Είναι μια πρόταση που εμείς υποστηρίζουμε ε, στεναρά και εργαζόμαστε σε 36 χώρες ε, συνεργασίας με έμφαση στις χώρες της ε, γειτονίας Ανατολικής και Νοτίου καλύπτουμε ένα σωρό διαστάσει και είναι τεράστιε σημασίε για μα. Επενδύουμε μαζί, φτιάχνουμε τοπικέ δυνατότητε ε, που μαζί και εργαζόμαστε σε θέματα βασικών πολιτικών επιτόπου. Είναι εταιρική σχέση για μα και θέλουμε να ε, συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτή τη συνεργασία και με το μέσο που σήμερα συζητάμε. Έχω να κάνω έξι παρατηρήσει. Ε, ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Ο συνάδελφο μόλι τον έφερε, θέλω να το επαναλάβω ότι το ΕΤΒΑ είναι παρόμοιο ε, και ε, τμήμα αυτής της προσέγγισης είναι ακριβώς ο συνδυασμός των διαφόρων μέσων που υπάρχουν ε, και αυτό θα αποδώσει για την εγγύηση που είναι νέο τις υπάρχουσες δυνατότητες blending που λειτουργούν πολύ καλά στον πρώτο πυλώνα Έχουμε τον δεύτερο πυλώνα και έπειτα το πολιτικό διάλογο και τις μεταρρυθμίσεις στην τρίτο πυλώνα. Εάν όλα αυτά γίνουν μαζί, και με όλους τους ε, μεμπλεκόμενους φορείς ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να υποδεχθεί πολύ ισχυρό και είναι πολύ χρήσιμο, ε, μια πολύ χρήσιμη εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη. Είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα στο πλαίσιο της BERD στις χώρες μας και πιστεύουμε πως πρόκειται για έναν πολύ δυνατό τρόπο να αποδώσουμε. Ελπίζουμε λοιπόν πως το Κοινοβούλιο θα προωθήσει κάθε μία από αυτές τις συνιστώσεις. Δεύτερη παρατήρηση, προσθετικότητα ξανά μανά. Ε, βασικός στόχος ε, της εγγύησης είναι να αυξηθεί το επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων για τις ε, επενδύσεις αυτές για να χρηματοδοτηθεί το χάσμα. Είναι τεράστιο αυτό το χάσμα και μόνο ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό. Άρα, και το είπαν άλλοι, ότι για να παροτρινθούν τα επίπεδα επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, η προσθετικότητα είναι πολύ βασική και δεν θα πρέπει αυτό να φοβήσει. Θα ήταν ε, ζημιογόνο κάτι τέτοιο. Παρακαλώ λοιπόν, το μήνυμά μας προς εσάς είναι μην διστάσετε να υψώσετε το πύχη και το επίπεδο ε, αποδείξεων που ζητάτε από μας τα επενδυτικά στους επενδυτικούς θεσμούς για να δείτε πώς αντιμετωπίζουμε τη συμφόρηση, ε, τα προβληματικά στοιχεία, ώστε να κινητοποιηθεί όσο γίνεται περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας. Πιέστε μας ε, και όχι μόνο θα πρέπει να μην βλάψουμε, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να παροτρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις ακόμα και σε χώρες που παλιότερα αυτό αποφευγόταν λόγω της αντίληψης περί κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ε, ενεργά να το περάσουμε στους ιδιώτες επενδυτές. Βασικός στόχος αυτής της εγγύσης δεν είναι να καλύψουμε το δικό μας κίνδυνο, τον, κίνδυνο δηλαδή των αναπτυξιακών χρηματοδοτικών ε, θεσμών, είναι να μπορέσουμε να περάσουμε και να συγκεντρώσουμε ιδιώτες και αυτό πρέπει να το πούμε ρητά. Τώρα, υπάρχει μια ολόκληρη σειρά φορέων που αναμειγνύονται εδώ, εμπλέκονται σε αυτή την, την πρωτοβουλία. Υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη για διάφορες περιφέρειες και πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε. Και πολλοί είστε εδώ σήμερα. Φυσικά και συνεργαζόμαστε πολύ στενά μεταξύ μας. Επίσης κάποιες φορές όμως ανταγωνιζόμαστε οι τους δε. Και αυτό συχνά είναι υγιές και έτσι η προσπάθεια για την εκπόνηση των καλύτερων δυνατών προτάσεων είναι διαρκής. Όμως θα πρέπει να διαχειριστούμε τα πάντα αμερόληπτα για να εξασφαλίσουμε ισότιμο πεδίο για όλους. Ε, θα πρέπει να το διαχειριστεί αυτό η Κομισιόν. ενθαρρύνουμε λοιπόν το Κοινοβούλιο να δώσει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της εγγύησης στην Κομισιόν, έτσι ώστε να εγγυηθούμε πως θα αναμειχθούν όλοι οι σωστοί φορείς και θα έχουν τις απαραίτητες εγγύσεις. Τώρα, οι λήψει αποφάσεων και η διακυβέρνηση. Είναι δημόσιο χρήμα και φυσικά χρειάζεται ο έλεγχος. Ο σχεδιασμός των δομών χρηματοδότησης και η ταχύτης είναι ζωτική σημασία αν θέλουμε να πείσουμε τους ιδιώτες επενδυτές να συνεργαστούν μαζί μας. Όλα τα ε, ε, οι, οι, εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούσαν να συμμετέχουν στα στρατηγικά διοικητικά συμβούλια για να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, αυτό θα εξασφαλίσει την παραπληρωματικότητα ανάμεσα στα όσα κάνουμε, όπως η πρωτοβουλία της ΕΤΕΠ για την ε, αντοχή, ε, πράγμα που καλύπτει κάποια είδη εγγύσεων. Τώρα, περισσότερα για το κλίμα. Εμείς πιστεύουμε πως ο στόχος για το κλίμα θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξος αν θέλουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας των Παρισίων. Οι ανάγκε για χρηματοδότηση για το κλίμα είναι τεράστιε, το ξέρουμε όλο αυτό και πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε στο άρθρο 8 να αυξήσουμε το στόχο στο 30% και αν όχι και παραπάνω. Ο ορισμό, κατά τη γνώμη μα, επίση είναι πολύ στενό για να είναι αποτελεσματικό. Το κλειδί για να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο είναι να μπορέσουμε να, να βάλουμε τη βιωσιμότητα στι αποφάσει περί δημοσίων επενδύσεων. Και έτσι γίνονται οι λαμβάνονται σωστέ αποφάσει και οι πράσινε επενδύσει απογειώνονται όταν υπάρχει όφελο για την επιχείρηση αλλά και χαμηλέ ε, εκπομπέ. Αυτό θα πρέπει να λοιπόν να συμπεριληφθεί στον ορισμό του άρθρου 8. Σημείο 6 και τελευταίο, Πρόεδρε, να διτηρήσουμε το ευρύ τον ορισμό των επενδύσεων. Εμείς από την πλευρά μας δουλεύουμε σκληρά, εξετάζοντας διάφορα επενδυτικά παράθυρα. Το να έχουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης μέσω συγκέντρωσης δομών, πρόθεση τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τοπική δανειοδότηση ώστε να μην είναι ευάλωτοι εταίροι που εκτίθεται σε κινδύνους ε, νομισματικών διακυμάνσεων, η εξασφάλιση προσιτής ε, και καθαρής ενέργειας. Υπάρχουν ένα σωρό ιδέες και ακόμη περισσότερες θα προκύψουν με το χρόνο, σε το χρόνο. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί γιατί η ανάγκη για τις χρηματοδοτικές λύσεις θα, αλλάξουν, θα αλλάξει στο μέλλον. Ευχαριστώ, σταματώ εδώ και με τα χαρά θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζόμς Και τώρα, όπως είπα κατά λάθος προηγουμένως, έχει το λόγο κύριος Παολούτσι, ειδικό ε, εκπρόσωπος Παγκόσμιας Τράπεζας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Βέλιο Λουξεμβούργο και στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία και σε μας να είμαστε παρόντες σήμερα. Μιλώ εξ ονόματος ε, της, ε, του ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας, Gold Bank Group, που ε, συμπεριλαμβάνει και ιδιώτες και το δημόσιο των διαφόρων κρατών. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, καλώς ορίζουμε και εμείς την πρωτοβουλία αυτή και ιδιαίτερα έχοντας υπόψη ότι μετά το 2015 και όλες τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην Αντίσα Μπέμπα, Νέα Υόρκη και Παρίσι, τώρα έχει έρθει η ώρα της υλοποίηση όλων αυτών. Της υλοποίηση των δεσμεύσεων και των στόχων που είναι φιλόδοξη πλην εφικτή. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης κινδυνεύουν όμως από την ε, ε, ε, ύπαρξη των σειράξεων. Το 2030 ο μισός πληθυσμός της γης θα ζει σε εύθραυστα κράτη. Γι' αυτό κατανοούμε για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικές ε, οι πρωτοβολίες σαν αυτή που συζητούμε σήμερα. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα για δράση και μάλιστα τώρα είναι αυτή η στιγμή. Ένας τρόπος ε, να αντιμετωπίσουμε θέματα υγείας, παιδείας, ε, να βγει ο κόσμος από τη φτώχεια και να αντιμετωπιστεί η εύθραυστη κατάσταση σε μια χώρα είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι εκ των όνου κάνευ. Μπορεί να μην είναι η πανάκια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο για να φεύγουν οι άνθρωποι από την ένδια. Εγώ μιλώ εξ ονόματος ενός ε, θεσμού που έχει ε, ως στόχο τον τερματισμό της απόλυτης ένδυας και την ενίσχυση του 40% του πληθυσμού της γης. Τα τελευταία 70 χρόνια έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά ε, σε αυτό το τομέα. Για να σας δώσω μια ιδέα, την τελευταία δεκαετία είχαμε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια υποστήριξη σε ευαίσθητα κράτη, εκ των οποίων 71 δις ε, για την ανάπτυξη του ιδιωτικού ε, τομέα. 9 δις σε ευαίσθητα έφθραυστα κράτη και 3 δις ε, σε θέματα αντίστοιχα που μας απασχολούν σήμερα. Έχουμε λοιπόν μια εμπειρία και βασιζόμενη σε αυτή και βασιζόμενη και στην ανάγκη να περάσουμε από τις δηλώσεις του 2015 επιτέλους σε δράση. Θεωρούμε ότι το ΕΤΒΑ είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ισχυρό εργαλείο για να αυξηθεί η, η ε, μόχλευση ε, υπάρχει επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια που πρέπει όμως να ενισχυθεί και από ιδιωτικούς πόρους και να γίνουν τα δισεκατομμύρια τρισεκατομμύρια. εκατομμύρια. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν οι θέσει απασχόληση εκείνε που χρειάζονται για να βγει ο κόσμος από τη φτώχεια. Είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετική σημασία να επενδύσουμε σε δημιουργικές αγορές. Πάνω από 70% των κρατών που μαστίζονται από ε, σειράξεις είναι ε, στο κατώτατο ε, όριο του καταλόγου της Παγκόσμιας Τράπεζας που λέγεται Doing Business. Αλλά ε, ακόμα και αν δημιουργήσουμε την αγορά δεν υπάρχει πανάκια, δεν υπάρχει μαγική λύση για να ε, ξεφύγει από την ένδυα ένα κράτος ή από τον κίνδυνο. Λάθη κάνουμε κι εμείς και μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αλλά η ανάπτυξη είναι και μια πολιτισμική διεργασία και χρειάζεται δεκαετίες. Και βρισκόμαστε εδώ για να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον. Δεν θα επιτύχουμε τα αποτελέσματα αν δεν είμαστε συγκεκριμένοι και ευστοχευμένοι σε αυτό που κάνουμε και να ξέρουμε ότι είναι μια προσπάθεια συλλογική. Είναι κρίσιμε οι εταιρικέ σχέσει. Δεν μπορεί κανένας από μόνος του. Επαναλαμβάνω, θα δεις, δεν γίνονται τρεις χωρίς μόχλευση των πόρων. Πόροι που υπάρχουν και πόροι που δημιουργούνται. Επιτρέψτε μου να επεκταθώ σε κάποια από τα σημεία. Πώς θα εμπλέξουμε τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε κάποιες αρχές για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Παγκόσμια Τράπεζα. Τι σημαίνει. Θα πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να επιτρέπεται να πηγαίνει πρώτος να επενδύσει στις αγορές. Όταν αισθάνεται και θεωρεί, και τι εννοώ ιδιωτικό τομέα, ε, ε, περιφερειακό, εθνικό, διεθνή. Όταν ο ιδιωτικός τομέας δεν βρίσκει εκείνες τις συνθήκες που θέλει για να επενδύσει σε μια χώρα ή ομάδα κρατών, τότε ερχόμαστε εμείς ως αναπτυξιακοί εταίροι ε, να συνεργαστούμε με τις χώρες για να δημιουργηθούν οι ε, προϋποθέσεις για να έρθουν ιδιωτικές επενδύσεις. Αν δεν επενδύει λοιπόν ο ιδιωτικό τομέα, ερχόμαστε εμεί ε, με χρηματοδότηση πάντα υπό όρους, για να υποστηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα. Είπαν και οι προλαλήσατε συνάδελφοι και τονίζω και πάλι την αρχή τη προσθετικότητα. Τι σημαίνει αυτό. Τι εννοούμε όταν λέμε προσθετικότητα και θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο blending. Το IFC για την προσθετικότητα τι σημαίνει. Όταν χρηματοδοτούμε τον ιδιωτικό τομέα ε, θα πρέπει να αποφύγουμε στρεβλώσεις της αγοράς, προβλήματα στην αγορά, αποτυχίες της αγοράς. Θα πρέπει να υπάρχει αηφορία, βιωσιμότητα και κυρίως διαφάνεια σε αυτή την προσπάθεια. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Έχει σημασία το ΕΤΒΑ να ευθυγραμμιστεί με τους άλλους δύο πυλώνες. Δηλαδή, το είπα και προηγουμένως, αν δεν μπορεί ο ιδιώτης να μπει σε μια αγορά, πρέπει εμείς να το βοηθήσουμε, να δημιουργήσουμε το πλαίσιο, το περιβάλλον με τεχνική βοήθεια, και ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας είναι κρίσιμοι. Αν δεν έχουμε αυτούς δεν πρόκειται να έρθει ο ιδιωτικό τομέα. Θα ρίχνετε λεφτά σε πρωτοβουλίε που είναι καταδικασμένες να αποτυγχάνουν. Και ένα τελευταίο. Εδώ γίνεται λόγος για επενδύσεις και πώς ε, εργαζόμαστε στις αγορές και συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας και να ενθυμούμαστε ότι τα έργα αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε μια πολύ γερή γνώση του τοπικού περιβάλλοντος. Δεν μπορείς από τις Βρυξέλλες να αποφασίζεις χωρίς να ξέρεις τι ε, ε, ισχύει και τι επικρατεί επιτόπου. Δηλαδή, όποιος και να εφαρμόσει αυτούς τους πόρους επιτόπου θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση και στενή σχέση με τις ε, χώριες αγορές, τους τοπικούς παράγοντες και εκείνους τους θεσμούς που λειτουργούν στις χώρες αυτές. Ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ε, προέλευσης. Αυτά ολοκληρώνω εδώ και σταματώ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Yes, thank you so much. So we have now a very broad uh, scheme. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα ιδεών. Τι θα πρέπει να κάνουμε, τι δεν θα πρέπει να κάνουμε. Και όπως ήθιστε θα δώσω το λόγο πρώτα στους εισηγητές οι κυρίες προηγούνται. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και σε αυτό το νέο πάνελ και τους ε, προσκεκλημένους μας για τις ε, εισηγήσεις τους. Είναι αλήθεια ότι ε, αυτό είναι που θέλουμε να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε με αυτό το κονδύλι, αυτό το ταμείο και τι όχι. Το θεωρητικό κομμάτι θα πρέπει να είναι πιο απλό αλλά να παραπέμπει άμεσα στον κανονισμό μας και ήταν περίπλοκο ο προπολογισμό γιατί αρκετοί ε, ομιλητέ αναφέρθηκαν στον τρίτο και στον ε, δεύτερο πυλώνα που είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντική με τον ίδιο τον ε, κανονισμό. Δηλαδή τον πρώτο πυλώνα. Εγώ έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με την συνεργασία των διαφορών θεσμών. Εσείς είπατε ότι κάποιες φορές ανταγωνίζεστε μεταξύ σας και ότι δεν είναι ο ανταγωνισμός, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε πως μια προστεθέμενη αξία αυτού του ταμείου θα είναι η απαραίτητη συνεργασία που θα πρέπει να συναυθεί ανάμεσα στι διάφορε επενδυτικέ και αναπτυξιακέ ε, τράπεζες και θεσμούς εσείς πώς βλέπετε ότι μπορεί να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία ανάμεσα στις τράπεζες και άλλη συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά τα παράθυρα τα επενδυτικά όπου είπατε ότι πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτός ο ορισμός, πιο χαλαρός και τουλάχιστον στη δική μας πρόταση ως εισηγητές δεν προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε τον ορισμό των παράθυρων των επενδυτικών γιατί μας φαίνεται ότι για την ώρα είναι αρκετά ευρύς αυτός ο ορισμός. Θα ήθελα να καταλάβω τι είδος, ε, γιατί είδος επενδυτικά παράθυρα μιλάμε. Μιλάμε για συγκεκριμένες χώρες, για συγκεκριμένα θέματα, για ε, συγκεκριμένους τομείς. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να ε, ορίσουμε αυτά τα επενδυτικά παράθυρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω βεβαίως διότι έχετε και εσείς μεγάλη εμπειρία με θέματα EFSI. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον συμβασμό EFSI, ποια πράγματα μπορούμε να πάρουμε και αυτομάτως να τα εντάξουμε στο νέο ταμείο EFSD. Θα, ε, είναι πολύ χρήσιμο να δούμε ε, ποια στοιχεία μπορούμε να περάσουμε ε, σχεδόν αυτούσια στο EFSD και ποια όχι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Τώρα ο κύριος Κούκαν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πλήρης επένων και ευχαριστειών. Όσα είπα για το πρώτο πάνελ τα αξίζει και το δεύτερο. Διότι κράτησε την συζήτηση σε πολύ ρεαλιστικό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης. Και κύριε Πρόεδρε θα πρέπει με μεγάλη σοβαρότητα να εξετάσουμε τι θα πρέπει να περιλάβουμε και τι θα πρέπει να αποφύγουμε να περιλάβουμε. Έχω δύο σύντομα ερωτήματα. Πώς βλέπετε από την οπτική των οργανισμών σας τη συνεργασία με άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς θεσμούς σε ό,τι αφορά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων του EFSD. Και δεύτερο, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Ποιες δυσκολίες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ε, προτάσεων αυτών, των μηχανισμών αυτών. Γιατί το θέμα αυτό είναι σημαντικό και ευαίσθητο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος ε, Φουρτουλίτσας. Ευχαριστώ. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι σήμερα συμμετείχα σε γεύμα εργασία με διμερείς οργανισμούς Χρηματοδότηση από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και οφείλω να πω ότι από την αρχή οι διμερείς αυτοί οι οργανισμοί χρηματοδότησης συμβάλλουν ενεργά στην διαμόρφωση νέας διευκόλυνσης για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Και μιας και έχουμε εδώ και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από αυτούς τους διμερείς οργανισμούς να παίξουν ορατό ρόλο στο σχεδιασμό τη συνεργασία αυτή. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμηση και Ανάπτυξη. Ίσως είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να λάβουμε κάποιε απαντήσεις. Ήδη ο συνάδελφός μου έθεσε το ερώτημα. Αυτοί οι 15 οργανισμοί πώ θα συνεργαστούν. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός. Εν τέλει, δε, θέλω να τονίσω και πάλι και να υπογραμμίσω ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το EFSD, αυτό το ΕΤΒΑ, e δεν θα επικαλυφθεί με υφιστάμενους μηχανισμούς και διευκολύνσεις και πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προσφέρουμε κάποια καινοτομία πιο εξελιγμένη με την αναγκαία ευκαμψία και ιδίω λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς ή μάλλον τις περιοχές ε, στις οποίες στοχεύουμε, δηλαδή Αφρική και χώρες της ε, Ανατολικής Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Και πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό για να προαχθεί η πραγματική προσθετικότητα και να προσελκυστούν ενδεχόμενοι ιδιώτες επενδυτές. Ευχαριστώ. Κύριε Τέιλορ. Τέλερ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ που οργανώσατε την ακρόαση. Ακούσαμε εκπροσώπους πολλών οργανισμών που μας εξήγησαν ποια πράγματα γίνονται. Πολύ χρήσιμο. Κάτι που εμένα, για μένα παραμένει κλειστό είναι τι θέλουμε να πετύχουμε με τον νέο αυτό μηχανισμό. ιδρύθηκε αυτός, όπως λέει, για να καταπολεμήσει τις αιτίε που οδηγούν πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις χώρες τους, διότι δεν τα βγάζουν πέρα εκεί, επί τόπου. Και θεωρούν ότι εδώ, στην Ευρώπη, αν φτάσουν, μπορεί να περάσουν καλύτερα. Παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν 350 εκατομμύρια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά 400 από την πολιτική γειτονία και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεω, τα οποία είχαν ήδη οριστεί. Δεν θα αλλάξει τίποτα υποτίθεται στην διαχείριση των ταμείων αυτών, αλλά προωθείται η προσπάθεια επίτευξη του στόχου, δηλαδή να δημιουργηθούν οι βάσει ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην εγκαταλείπουν τι χώρε του. Προ δύο εβδομάδων, αντιπροσωπεία τη Επιτροπή Αναπτύξεω πήγε σε μια χώρα που δεν βρίσκεται βέβαια στην αιστεία τώρα, στο Τσάντ, δηλαδή στο στόχο σα, και είδαμε εκεί ποιε είναι οι αιτίε τη μετανάστευση, οι ποιε μπορεί να είναι. Και το πρώτο ήταν ότι τα κρατικά έσοδα της χώρας αυτής, του Τσάντ, μειώνονται σημαντικά, μαζικά. Γιατί, Γιατί η μοναδική, ο μοναδικός πόρος συναλλάγματος για το Τσάντ ήταν τα κοιτάσματα πετρελαίου, το οποίο, τα οποία όμως εκχωρήθηκαν σε διεθνή σύμπραξη με έδρα την Ελβετία. Το Τσάντ στη σύναψη της συμβάσεως αυτής έλαβε προκαταβολή από τα αναμενόμενα κέρδη από την πώληση του πετρελαίου. Τώρα όμως μειώθηκε η τιμή του πετρελαίου και τα αναμενόμενα κέρδη της εταιρείας αυτής, Lemcor, δεν ανταποκρίνονται πλέον στα όσα συμβατικά είχε υπογράψει και τώρα το Τσάντ καλείται να συμπληρώσει τα ελλείμματα. Από την τσέπη του το Τσάντ, που αυτό σημαίνει ότι τα κρατικά έσοδα δεν αρκούν πλέον για τα υπόλοιπα παιδεία, υγεία και ούτω καθεξής. Δεύτερο, προδιετίας. 25.000 πολίτες του Τσάντ επέστρεψαν στο Τσάντ από την κεντροαφρικανική δημοκρατία λόγω συγκρούσεων που γίνονται εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν κάποιο εισόδημα εκεί και καλές θέσεις στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Εδώ και δύο χρόνια περιμένουν μέσα σε άθλιες συνθήκες, σε στρατόπεδα του Τσάντ, αναμένουν από το, κέντρο, από το κράτος του Τσάντ να τους αναγνωρίσει ως πολίτες του και να τους χορηγήσει τα κατάλληλα έγγραφα ώστε να μπορέσουν να βρουν δουλειά στο Τσάντ. Και τρίτο παράδειγμα, γιατί μπορώ να σας πω και άλλα πολλά, χρηματοδοτούμε στο Τσάντ ένα σύστημα προστασίας συνόρων με 12 ε, σταθμούς και με σκάφη τα οποία περιπολούν στον ποταμό με συνέπεια οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή του Τσάντ που μέχρι τώρα πήγαιναν τα βόδια τους στην ε, βορειοανατολική Νιγηρία για να τα πουλήσουν εκεί, τώρα δεν έχουν πρόσβαση πλέον στην βορειοανατολική Νιγηρία. Και βεβαίως διαμαρτύρονται, διότι αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην οικονομική του δραστηριότητα. Αυτά είναι τα προβλήματα. τα οποία τα φτιάξαμε εμεί, τα προκαλέσαμε εμείς. Και με αυτά τα γελία 57 εκατομμύρια πώς θα αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τις αιτίε αυτές και να μην προσπαθούμε και πάλι να δημιουργήσουμε κάποιου μηχανισμούς πλατσέβο. Ευχαριστώ. Είπαμε δύο λεπτά, ε. Η κυρία Χαουτάλα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είμαι πεπισμένη ότι για να στηθεί ένα ταμείο όπως το ΕΤΒΑ χρειάζεται πραγματογνωμοσύνη και συμβουλές τις οποίες θέλουμε και στις οποίες ε, προστρέχουμε. Είπατε κάτι σημαντικό μεταξύ άλλων. Αυτό είναι η γνώση και η παρουσία της εγχώριας πραγματικότητας για να μπορεί να έχει αντίκτυπο αυτή η προσπάθεια και να πιάνουν τόπο. Και θέλω να σας ρωτήσω στα πλαίσια ε, ε, του υγιούς ανταγωνισμού και της άμυλας, ποιος έχει την καλύτερη παρουσία από εσά σε χώρες υποσαχάριας Αφρικής. Ή για αυτό που σας ανέφερε ε, ο κύριος Τσέλερ μόλις, ποιος έχει την καλύτερη γνώση της τοπικής πραγματικότητας. Δεν έχει ζητήσει κανένας άλλος το λόγο. Δύο λεπτά έκαστος για να απαντήσετε, παρακαλώ να τα τηρήσετε, γιατί ε, πεντέμιση θα πρέπει να έχουμε τελειώσει. Ποιος θέλει το λόγο, παρακαλώ very quickly to stay within two minutes. First question was on cooperation. How does cooperation work among institutions? I think it's a very... Καταρχάς για τη συνεργασία μεταξύ των θεσμών. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και μεγάλη πρόκληση, διότι πρόκειται για εγγυήσει που πρέπει να μοιράζονται ανάμεσα στι διάφορε τράπεζε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σαφής, μια σαφή χαρτογράφηση των κινδύνων με κοινή αξιολόγηση κινδύνων τη ίδια εγγύηση. Διαφορετικά δεν λειτουργεί. Άμα η μία τράπεζα λέει εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω έχει τον τάδε κίνδυνο, ενώ η άλλη τράπεζα λέει τρία μείον, ε, μείον τρία μάλλον, ε, κίνδυνο, ε, δεν θα συνεννοηθούμε. Επίση είναι σημαντικό να έχουμε ε, ένα σαφές σύστημα ε, μέτρησης αντικτύπου, γιατί πάλι το ίδιο θα συμβεί αν ένας λέει το ένα και ο άλλος το άλλο. θα πρέπει να μπορούμε να, να, να τα μετρήσουμε όλα αυτά. Και τέλος, η συνεργασία ε, φυσικά βασίζεται στη συνεργα... στην εμπιστοσύνη και σε κοινού στόχους. Τώρα, ε, ε σε, σε αντίθεση με το κλειστό σύστημα ε, επενδύσεων. Καταρχάς η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει ε, τη γνώμη της σε αυτό το σημείο. Σημαντικό είναι η γεωγραφική στόχευση, για παράδειγμα ευαίσθητα, ευάλωτα κράτη και εκεί να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί για τα θέματα, για το τομεί, γιατί είναι πολύ δύσκολο εκεί να βρούμε ιδιώτες. Ε, ε, ταυτόχρονα οι πιο προηγούμενε χώρες εταίροι μπορεί να βρίσκουν τις συγκεκριμένου τομείς που θεωρούν ότι είναι σημαντικοί ε, για θέματα πολιτικής. Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα από το ΕΦΣΥ. Θα πρέπει να βασιστούμε στο τρόπο λειτουργίας, γιατί χρησιμοποιούμε τη μέτρηση αποτελεσμάτων με το ΙΡΕΜ ε, και με το ε, Μηχανισμό Σταθερότητας, δηλαδή και με το BERD, ε, με τον ίδιο τρόπο μέτρησης δηλαδή. Είναι πολλά ερωτήματα για δύο λεπτά. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό Α, ναι, αυτό που δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από τα είναι οι πολιτικές ε, ε, κινδύνου της ε, ΕΤΕΠ. Εμείς θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο επικίσιους προς το κίνδυνο, δεδομένων των στόχων αυτού εδώ του προγράμματος. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να είναι πολύ στερεό πλαίσιο. Γιατί επιτόπου παρουσία, γιατί πρόκειται εδώ για διαγωνισμό ομορφιά. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις αντιπροσωπείε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ε, τους δικούς μας εκπροσώπους επιτόπου στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που διευκολύνει το γεγονός ότι αυτές οι αντιπροσωπείες ξέρουν ακριβώς ποιες είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην εκάστοτε χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος ε, Άντρισεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εφόσον εγώ αντιπροσωπεύω μια ομάδα 15 ε, φορέων, ξέρουμε πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε και να συνεργαστούμε ταυτόχρονα. Η χρηστή συνεργασία ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σημαίνει καταρχάς ένα ισότιμο ε, πεδίο και κοινέ προδιαγραφές για την εργασία που κάνουμε με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν 15 διαφορετικά σύνολα κανόνων όταν ε, συζητάμε για επενδύσεις και δεν χρειάζεται παρά μόνο μία φορά το χρόνο να συνεδριάζουμε για να εγκρίνουμε τις ε, αποφάσεις, τις επενδύσεις, να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτά τα project πρέπει να χρηματοδοτηθούν όταν πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Αυτό είναι η εμπειρία μας. Έχουμε αρκετά επιτυχίες δε επιτυχή προγράμματα στις χώρες ΑΚΕ για το κλίμα, όπου οι 15 μαζί με την ε, ΕΤΕΠ και το Αναπτυξιακό Ταμείο βρήκαμε κοινού κανόνε και κοινού τρόπους λειτουργία και εμπειρία μα εκεί νομίζω θα είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώ θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μα στο μέλλον. Για το ΕΤΒΑ και το σχέδιο των 15 ε, ευρωπαϊκών δημερών θεσμών είναι να κάνουν το πρώτο βήμα υποβάλλοντας κάποιες προτάσεις για κοινά προγράμματα, για συμπράξει συμπράξεις, κοινοπραξίες. Να το έχουμε δηλαδή δηλημένο το θέμα της συνεργασίας από τις προτάσεις που θα υποβάλουμε. Επίσης με διμερείς ε, ε, συμπράξεις ή συνεργασίες εκεί που υπάρχουν, υπάρχει ειδική εμπειρία, ειδικέ ιδέες και τέλος, νομίζω ανέφερα και νωρίτερα όσον αφορά την εμπειρία επιτόπου στις χώρες που στοχεύουμε, έχοντας το 1 τρίτο των χαρτοφυλακίων μας περίπου στην υποσαχάρια Αφρική και σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, δηλαδή πάνω από χίλια project, καταλαβαίνουμε, πιστεύω, έχουμε αρκετά καλή γνώση της αγοράς αυτής. Ευχαριστώ κύριε Ζώνς. Ευχαριστώ πολύ. Ένα γενικό σχόλιο μόνο. Σε σχέση με κάτι που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνώ. Εν είναι τεράστια τα προβλήματα και δεν είναι πανάκια η λύση και το ταμείο αυτό για τα πάντα. Κάποια προβλήματα θα λύσει, όχι όλα. Υπάρχουν ε, κάποια έργα που χρηματοδοτούνται μόνο με επιχορηγήσεις, με δοτήση, όχι με δάνεια. Αυτό είναι το γενικό σχόλιο. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ε, σε μεγάλο βαθμό. Τι είναι οι εγγύσεις. Όπως είπε και ο συνάδελφος από την ΕΤΕΠ στην απάντησή του, όταν μπαίνει στο θέμα των εγγύσεων, είναι πολύ ευαίσθητο τραπεζικό ζήτημα αυτό και οι τράπεζες είναι πάρα πολύ εχέμηθες και μυστικοπαθείς ως προς τις εξηγήσεις τους και τις προφορίες. Είναι δύσκολο να τις ε, εκμεύσεις. Ο καλύτερος τρόπος είναι να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των εγγύσεων. Και εδώ επανερχόμαστε σε αυτή την έννοια των ε, ίσων όρων παιχνιδιού. Πώς συνεργαζόμαστε. Ε, μην κάνετε επικαλύψεις, συνεργαστείτε. Ε, ε, είναι η αρχή και το κάνουμε αυτό. Και πάντα είναι περίπλοκο. Δεν υπάρχει απλός τρόπος να γίνει κάτι τέτοιο. Κάθε μέρα πρέπει να το εφευρίσκουμε από την αρχή. Με ενημέρωση, με ανταλλαγή πληροφοριών, με συμμετοχή σε μεγάλες συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Το είπα και προηγουμένως να συμμετέχουν και άλλοι ε, στρατηγικό επίπεδο, ας Και αν δούμε ότι υπάρχει ζήτημα να το πούμε. Ελπίζω ε, αυτό να ε, εισακουστεί. Ένα άλλο πολύ σημαντικό. Το ΕΤΒΑ δεν έχει να κάνει μόνο με τις εγγύησεις, αλλά με τα ρυθμίσεις στην πολιτική και τεχνική βοήθεια. Θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και το κάνουμε ήδη πολλοί από εμά εδώ, σε, πολλές, σε πολλά επίπεδα και ε, τα ιδρύματα στα οποία εργαζόμαστε και οι θεσμοί συνεργάζονται. Και όταν συνδυάζεται μια επένδυση με μεταρρύθμιση πολιτική, θα πρέπει να υποστηρίζεται αυτό και από ε, κάποιον άλλο θεσμό. Το θέμα δεν είναι μόνο να μην ανταγωνιζόμαστε για την επένδυση, αλλά να υποστηρίζουμε και τις μεταρρυθμίσει που γίνονται και να μην έχουμε ανταγωνιστικό ρόλο. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, για τι επενδυτικέ ευκαιρίε, τα παράθυρα. <coughs> Το κάνουμε αυτό και ε, στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και της Νότιας και ψάχνουμε επενδυτικές ευκαιρίες Τι γίνεται ας πούμε σε επίπεδο ε, το τοπικό νόμισμα ή ε, χρηματοδότηση μικρομεσαίων ή βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις ε, και φυσικά η ε, παρουσία οι χώρες, όλες τις χώρες που επενδύουμε έχουμε βαθιά γνώση του πεδίου βαθιά γνώση των κλάδων ε, με εμπειρογνώμονες και σε τραπεζικό τομέα. Πραγματικά, τομέα κλάδο, έχουμε παρουσία και κλάδο της επιχειρηματικής ζωής ε, παντού όπου επενδύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος, αλλά βεβαίω όχι λιγότερο σημαντικό, ο κύριος Παολούτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σύντομο, γιατί ήδη καλύφθηκα σε σημαντικό βαθμό από τον συνάδελφό μου κύριο Τζονς Κάποιοι θεωρούν ότι δεν συνεργαζόμαστε, όμως συνεργαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό και να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο λόγω του μεγέθους των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και λόγω του γεγονότος ότι πρέπει να καταδείξουμε ακόμη περισσότερο με την παρούσα πρωτοβουλία ότι προσφέρει value for money, ότι αξίζει δηλαδή. Και με υγιή ανταγωνισμό. Έχουμε στο δεύτερο που είπε ο William Jones και το υποστηρίζω, η παρουσία στο στρατηγικό ε, αυτό συμβούλιο ε, έστω και με καθώς παρατηρητού είναι σημαντική και θα είναι πολύ χρήσιμη. Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, ο κύριος Κούκαν ρώτησε ποιες είναι οι, ε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τους επενδυτές. Απουσία αγορών. Μιλούμε για ορισμένες χώρες που δεν έχουν αγορά. Μεγάλος κίνδυνος και αυτό οδηγεί στο δεύτερο σημείο. Θεσμοί δηλαδή που έχουν αποτύχει. Είχαμε κάνει μελέτη προετών που έδειξε ότι για να είναι μια χώρα στέρεα, με στέρεους θεσμούς, μπορεί να τις πάρει και 70 χρόνια. πάλι επανέρχομαι σε κάτι που είπε ο Τζόνς. Δεν είμαι ο καταλληλότερος. Ω εκπρόσωπο οργανισμού που δεν είναι Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Όμω, η στόχευση πρέπει να γίνει στους τομείς και στα προϊόντα και ως στους ίδιους τους θεσμούς. Για να σφυριλατήσετε μια καινοτόμα νοοτροπία, μια νοοτροπία δηλαδή που να στηρίζει καινοτομίες και να προσφέρει νέες λύσεις για καμιά φορά πολύ ε, ανυπέρβλητα προβλήματα. Ο οργανισμός μας έχει περίπου 20.000 μέλη προσωπικού και είμαστε παρόντες σε όλες τις αφρικανικές χώρες, με τα γραφεία μας στις αφρικανικές χώρες και στο AIDA Replenishment μία από τις δεσμές που αναλάβαμε ήταν να ενισχύσουμε την παρουσία μας σε έφραστες χώρες με πρόσληψη προσωπικού της τάξης των 200 μελών για την παρουσία μας στις έφραστες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε τους τρεις εισηγητάς, οι οποίοι θα κάνουν τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ένα λεπτό για τον κύριο Κούκαν. κάποια σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μιας και, μια και μας μένουν πέντε λεπτά, ποιος θέλει από εσά να μιλήσει. Πόσα είπατε, πέντε λεπτά. <laughs> Ένα λεπτό, για τον καθένα από εσά λέει ο πρόεδρο. Καλά, θα είμαστε σύντομοι, διότι η προσέγγιση μα είναι πολύ όμοια με αυτή του πάνελ. Ευχαριστώ που μιλήσατε για τους τρει πυλώνες, την διάδραση και την προσθετικότητα. Ο σχεδιασμό του EFST βασίζεται στην από μακρού χρόνου συνεργασία που έχουμε με έναν αριθμό ε, χρηματοδοτικών οργανισμών και από αυτούς που εκπροσωπούνται στο πάνελ αλλά και ε, των διμερών οργανισμών που μνημονεύτηκαν σήμερα. Μιλώ και για την Αφρικανική Τράπεζα Αναπτύξεως ως ε, ο ένας εκπρόσωπος που λείπει από το πάνελ σήμερα και για το σημαντικό ρόλο βέβαια των μη κρατικών οργανισμών που επίσης πρέπει να τονιστεί. Όλα αυτά δείχνουν ότι πραγματικά ε, είμαστε ισότιμοι, είμαστε στο ίδιο ύψος, ας το πω έτσι, ε, μεταξύ μας και ε, όλοι συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς τώρα. Πολύ σύντομα. Έχουμε πραγματικά πολύ ισχυρούς συνομιλητές και θεσμούς εταίρους. Πολύ σημαντικό διότι μιλούμε για 70 αφρικανικές χώρες της αφρικανικής γειτονίας με πολύ μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα και ίσως ορισμένοι να μην αντιλαμβάνονται ότι ένας από τους πιο δύσκολους στόχους είναι να βρεθούν ε, κατάλληλα έργα, project, που να μπορούν να χρηματοδοτηθούν, αλλά και που να σέβονται τις βασικές αρχές τις οποίες αναφερθήκαμε ήδη. Άρα είναι δύσκολο το καθήκον αυτό. Επαφιέμεθα στην ικανότητα των τραπεζών ε, να υλοποιήσουν τα έργα αυτά και γι' αυτό είναι κέρια σημασίας να έχουμε μεγάλο αριθμό συνομιλητών και εταίρων και θεσμούς οι οποίοι να μπορούν να υλοποιήσουν το πράγματι πολύ δυσχερές αυτό έργο. Τελευταίος εσείς. Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Εγώ έχω να πω ότι η είπατε εκπρόσωπος κυρία Μόγκερίνη η οποία έχει πρωταγωνιστήσει για αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμη ανάπτυξη. θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ένα μέρος αυτής της ε, συνεργασίας της ε, συνεταιρικής προσέγγισης με συμμετοχή όλων των φορέων, ώστε και οι ανάγκες των χωρών εταίρων, αλλά και η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλει μια συνολική προσφορά που να βασίζεται στα ισχυρά σημεία όλων μας. Γι' αυτό αυτό που είδαμε σήμερα με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων των διαφόρων άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών που ε, έχουν σχέση με τις χώρε μέλη μας και ο ρόλος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και όλων των αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου νομίζω ότι αποτελούν εν τέλει το σωστό μείγμα και σε ό,τι αφορά την εμπειρογνωμοσύνη και σε ό,τι αφορά την παρουσία επιτόπου. Όλοι από αυτούς έχουν κάποια ισχυρά σημεία, κάποια ισχυρότερα από άλλου και για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι το εργαλείο αυτό θα αποτελέσει πράγματι μια καινοτόμα προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ τα μέλη του πάνελ για τις χρήσιμες συμβουλές, ευχαριστώ τους Πρόεδρους Επιτροπών που προσήλθαν και ήταν παρόντες σήμερα και σας υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνάντησή μας θα διεξαχθεί στις 21 Τρίτου στις 5.30 όπου οι εισηγητές να παρουσιάσουν επισήμως το σχέδιο εκθέσεως. Ευχαριστώ επίσης που προσήλθατε και που μας δίνετε την ευκαιρία έτσι να προχωρήσουμε στο σωστό δρόμο. Και καλό σας βράδυ.